Καλημέρα σε όλους. Παρακαλώ καθίστε, διότι θα ξεκινήσει η συνεδρίαση. Κύριε Ρωμέβα, παρακαλώ καθίστε. How are you? Did you have a good time? Good.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 Παρακαλώ, καθίστε. Καλημέρα λοιπόν σε όλους και πάλι. Ελπίζω να περάσατε καλές διακοπές όλοι σας και να έχουμε επιστρέψει πιο χαλαροί και πιο ξεκούραστοι για να συνεχίσουμε τις εργασίες μας πλέον. Καταρχάς, στην ημερήσια διάταξη σήμερα έχουμε την έγκριση της ημερήσια διάταξη. Να σας πω ότι το σημείο υπαριθμών 8 της ημερήσια διάταξη, στο οποίο η κυρία Ιώτοβα θα μας έκανε μία παρουσίαση της ε, αντιπροσωπείας που μετέβει στη Βουλγαρία. Η κυρία Ιώτοβα δεν μπορεί να παραστεί σήμερα, επομένως ε, αναβάλλεται το συγκεκριμένο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Να σας πω όμως ότι η Γραμματεία έχει ήδη ετοιμάσει μία σύντομη έκθεση της επίσκεψης αυτής της αντιπροσωπείας, η οποία θα διανεμωθεί σε όλους σας. Η κυρία Πατραονέβες. Πρόεδρε, θα ήθελα να προτείνω το σημείο 10 της σημερινής διάταξης να εξεταστεί αμέσως μετά τις ψηφοφορίες ή δυνατόν. Το 10 σημείο, λέω, θα ήθελα, αν γίνεται, να το εξετάσουμε αμέσως μετά τις ε, ψηφοφορίες. Ε, αν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Πρόεδρε, σε σχέση με το σχέδιο ημερήσιας διάταξης που λάβαμε, πιστεύω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε σχέση με την πρόταση της κυρίας Πατράου Νέβες πιο συγκεκριμένα. Αυτό το σημείο 10 κανονικά θα πρέπει να είναι μετά την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 12 και 13 Ιουλίου. Γιατί έχουμε και τα πορίσματα εκεί της συνεδρίασης των συντονιστών. Ε, και αυτά θα τα εξετάσουμε στο σημείο 10. Οπότε, γιατί να εγκρίνουμε τα πρακτικά όπου υπάρχουν τα πορίσματα της συνεδρίας των συντονιστών που θα εξετάσουμε όμως ε, στο σημείο 10. Θα πρέπει να αλλάξει η σειρά δεν μπορούμε να εγκρίνουμε τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης ε, πρωτού συζητήσουμε και αποφασίσουμε αυτά που προβλέπονται στο σημείο 10. Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λογικό να ακολουθήσουμε άλλη πορεία. Στο σημείο 10 θα συζητήσουμε αυτά τα πορίσματα της συνεδρίας των συντονιστών. Οπότε δεν μπορούμε ε, να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας για την έγκριση των πρακτικών βάσει του σημείο 2. Ξαναλέω, σε παράρτημα ε, στο σημείο 10 υπάρχουν τα πορίσματα συνεδρίας των συντονιστών. Έχετε δίκιο σας, καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι πάντα τα πρακτικά θεωρούνται ότι εγκρίνονται στο πέρας της συνεδρίασης εάν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση. Έχετε δίκιο, εν γέννη πάντα εδώ στην Επιτροπή Αλληλείας τα πρακτικά εγκρίνονται στο τέλος της συνεδρίασης εάν και εφόσον δεν έχει παρουσιαστεί κάποια ένσταση. Γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να αλλάξουμε το σημείο στην ημερήσια διάταξη και ανάλογα θα εγκριθούν και τα πρακτικά. Μάλιστα, είναι η τρέχουσα πρακτική. Δηλαδή, αν δεν προκύψουν ενστάσεις και συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχουν προκύψει ενστάσεις, Ωραία, εγώ θεωρώ ότι τα πρακτικά θα πρέπει να εγκριθούν μόλις διευκρινιστούν όλα τα σημεία υπό το σημείο 10. Ε, τι να σας πω, θεωρώ ότι το να εγκρίνουμε κάτι που δεν έχουμε συζητήσει δεν είναι η ενδεδειγμένο, ο ενδεδειγμένος τρόπος εργασίας. Ε, έχουμε το σημείο 1 συγκεκριμένα στα πορίσματα της συνεδρίασης των συντονιστών ε, και εκεί το περιεχόμενο μπορεί να τροποποιηθεί μετά τη συζήτηση. Ε, δεν μπορούμε άρα να θεωρήσουμε τα πρακτικά εγκεκριμένα. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν γίνεται να εγκρίνουμε πρακτικά προηγούμενε συνεδρίε προτού τα συζητήσουμε. Eh, eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να πω Πρώτον, ε, να, ε, δεν θα ήθελα να διαταράξω τη σειρά των συζητήσεων ε, λόγω τη ημερήσια διάταξη. Δεύτερον, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Α ακολουθήσουμε όποια σειρά θέλουμε. Τρίτον, τα πρακτικά είναι αυτά που είναι. Έγιναν κάποια πράγματα, δεν θα γράψουμε ιστορία τώρα. Καλούμεθα να εγκρίνουμε τα πρακτικά, αλλά δεν θα γράψουμε ιστορία, ξαναλέω. Τι σχέση έχει η έγκριση των πρακτικών με τις αποφάσεις των συντονιστών. Ε, ας κάνετε ό,τι θέλετε. Ε, δεν θέλω εγώ τώρα για ένα θέμα ίσονος σημασία να δημιουργήσω πρόβλημα ε, λόγω της σειράς των υποσημείων της ημερήσιας διάταξης. Αυτά που συνέβησαν, συνέβησαν. Ποιος θα τα αμφισβητήσει, θα πούμε εμείς ότι δεν συνέβησαν. Ε, ε, δεν μπορούμε να τοποιήσουμε τις αποφάσεις αφού ε, αυτή στιγμή έχει συμβεί κάτι. δεν μπορούσα παρά να το πω αυτό, συγγνώμη. Δεν υπάρχει λόγος. Μπορούμε να εγκρίνουμε τα πρακτικά στην επόμενη συνεδρίαση και επομένως λύθηκε το πρόβλημα. Ωραία. Να με αυτό ολοκληρώσαμε τα σημεία 1 και 2. Λαμβάνοντα υπόψη το αίτημα τη κυρία Πατράουνα Νέβε, τη κυρία Ιώτοβε και το γεγονό ότι θα εγκρίνουμε τα πρακτικά στην επόμενη συνεδρίαση για να μην υπάρχει πρόβλημα, εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Επομένω, επειδή δεν υπάρχει αντίρρηση, θεωρούμε ότι εγκρίνεται. Περνάμε στο σημείο παριθμών 3 τη ημερήσια διάταξη, λοιπόν, οι ανακοινώσει τη Προέδρου. Θα ήθελα να σα πω ότι η ομάδα των φιλελευθέρων μου απέστειλε μια επιστολή όπου ανακοίνωνε την αντικατάσταση της κυρίας Μπρίτα Ρέιμερς από τον κύριο Χατζημαρκάκη ως τακτικό μέλος της Επιτροπής μας. Η απόφαση θα επικυρωθεί στην επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας, η οποία θα πρέπει να επιβεβαιώσει τη συγκεκριμένη αλλαγή. Να ευχηθούμε στην κυρία Ρέιμερς ό,τι καλύτερο στη ανέα της καθήκοντα σήμερα θα είναι εδώ διότι είναι εισηγήτρια για τον προϋπολογισμό και την ευχαριστούμε για τα όσα έκανε στα πρώτα αυτά δυόμιση χρόνια ε, εντολής που είχαμε. Ωραία, σας ευχαριστώ και να περάσουμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 4 της ημερήσιας διάταξης, ε, ψηφοφορία για την ε, αλληλευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη Συμφωνία Αλληλευτικής Έμπραξης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Πράσινου Εκροτηρίου. Η εισηγητής είναι ο κύριος Γκάλακερ, έχουμε συζητήσει το θέμα επανειλημμένος, είχαμε γνωμοδετήσει από την Επιτροπή Ανάπτυξης και την Επιτροπή προπολογισμών. Η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών ήταν 20 Ιουνίου, δεν παρουσιάστηκε καμία τροπολογία. Να ολοκληρώσω και θα σας δώσω το λόγο. Η διαδικασία, όπως γνωρίζετε, είναι βάση του άρθρου 43.2 των συνθήκων και του άρθρου 218.6α να δώσω το λόγο στον κύριο Φερέιρα που έχει ζητήσει το λόγο και μετά θα δώσουμε το λόγο στον εισηγητή. Ο κύριος Φερέιρα. Ζητώ συγγνώμη Πρόεδρε, ζήτησα το λόγο πρωτού μπείτε σε αυτό το σημείο αλλά δεν με είδατε. Ζητώ συγγνώμη που σα διέκοψα, συγγνώμη για τη σύγχυση. Θέλω να αναφερθώ πάλι στο προηγούμενο σημείο. Ε, ήθελα να θυμίσω εδώ ότι υπήρχε η ευκαιρία με άλλους δύο συναδέλφους από τους συντονιστές των Σοσιαλιστών ε, και των Πρασίνων να στείλουμε στη Γραμματεία και στην ε, Επιτροπή μία επιστολή όπου προτείναμε να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη σημερινή σημερινής ένα υποσημείο ε, σχετικά με την ε, κατανομή των εκθέσεων για την κοινή αλληλευτική πολιτική. Πλην όμως δεν συμπεριλήφθηκε αυτό το σημείο και ήθελα απλώς να το θυμίσω. όλοι οι συνάδελφοι έχουν πρόσβαση σε αυτή την επιστολή με το αίτημά μας και όπως έγινε η συζήτηση για αυτό το θέμα στη συνεδρία των συντονιστών, αντιλαμβανόμαστε ότι θα ήταν καλύτερο για όλους, καλύτερο για τις εργασίες της Επιτροπής μας να έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτό το σημείο κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης της Επιτροπής Αλίας. Ε, εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι καλύτερο έτσι και λυπάμαι που δεν συμπεριλήφθη το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη. Ε, σε αυτή τη συνεδρίαση, αν έχουμε χρόνο, καλό θα ήταν να συζητηθεί ή στην επόμενη συνεδρίαση. Ε, Ήθελα μόνο να επενθυμίσω το αίτημά μας αυτό. Eh, Ωραία, θα το δούμε αυτό στο τέλος. Εγώ προσωπικώς, εσείς βεβαίως μπορείτε να έχετε και την άποψή σας, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί πρώτα στους συντονιστές και μετά να περάσει στην Ολομέλεια της Επιτροπής μας. Εάν όμως εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να συζητηθεί πρώτα εδώ, στην Επιτροπή, πολύ καλά θα το συζητήσουμε ή στο τέλος συνεδρίασης ή στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Ελίας. Εξακολουθώ να θεωρώ όμως ότι είναι πρώτα αρμοδιότητα των συντονιστών και εάν θέλετε καλό θα ήταν στην επόμενη συνεδρίαση να ε, τα δούμε τις επιστολές και να λάβουμε και τη σχετική απόφαση. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Γκάλαγκερ για να μας ε, πει ε, τα του θέματος που μας απασχολεί και αν δεν θέλει να μιλήσει θα περάσουμε απευθείας στην ψηφοφορία. Θέλετε το λόγο? Ναι, παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έγιναν ε, διάφορε ανταλλαγέ ε, απόψεων για αυτή την έκθεση που δεν είναι αμφιλεγόμενη. Αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα να δούμε ποιε είναι οι επιπτώσει όλων αυτών. έχω αναφερθεί σε αυτό γενικά σε προηγούμενε συνεδριάσει σήμερα εκπνέει το προηγούμενο πρωτόκολλο ε, και μετά από 4,5 χρόνια εφαρμογής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε διαπραγματεύσεις για ένα νέο πρωτόκολλο το ε, Δεκέμβρη του 2010 και από Σεπτεμβρίου 2011 θα αρχίσει να ισχύει το νέο πρωτόκολλο για μια τριετή περίοδο. Το Συμβούλιο κατέληξε ε, σε συμπεράσματα, αλλά χρειάζεται η πρώτερη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου, ούτως ώστε να συνεχίσει η αλληλεία ε, στα ύδατα του Πράσινου Ακροτήριου και είναι απαραίτητο ε, να εγκριθεί προσωρινά το νέο πρωτόκολλο βάσει του άρθρου 15. Η άποψή μου είναι ότι μπορεί να θεωρηθεί αυτό, ε, αυτή η χώρα ε, ως, αυτή που έχει, ε, ως ότι είναι μεταξύ αυτών που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις στην Αφρική και η αλληλευτική πόρη δεν είναι τόσο σημαντική αλλά συμπεριλαμβάνουν εμπορικά σημαντικά είδη ψαριών έχουμε μικρά πελαγικά είδη, τόνους, κάποια βενθικά είδη, αστακούς φυσικά ε, και ε, έχουν αρθεί οι φράγμοι για την πρόσβαση στις ευρωπαϊκές ε, αγορές για τα είδη αυτά και η χώρα είναι μέλος της ΕΚΑΤ. Επίσης υπάρχουν συμφωνίες με την Ινδία και με την Κίνα, αλλά τέλος πάντων η σημαντικότερη διμερή συμφωνία της χώρας αυτής είναι αυτή που έχει συναυθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα λιεύματα των τόνων από ευρωπαϊκά σκάφη ανέρχονται ή μάλλον δεν ξεπερνούν το 0,2% των αλλιευμάτων από τα συγκεκριμένα ε, αλλιευτικά είδη. Δεν είναι τόσο σημαντικά λοιπόν. Και ε, η τον αλλιευτική δραστηριότητα είναι ίσονο σημασία. Ε, σχετικά τώρα με είδη καρχαριών όπως ο μπλε καρχαρίας δεν οδηγεί σε ε, εξάντληση των ε, αποθεμάτων. Βέβαια, βέβαια υπάρχει και μία μικρή αβεβαιότητα σε σχέση με την εκτίμηση της κατάστασης των αλλιευμάτων. Όπως είπαν οι συνάδελφοι που ήταν εκεί, ε, μας είπαν ότι οι επιστήμονες παρακολουθούν και συμμορφώνονται με τις επιστημονικές συμβουλές της και κυρίως για την αλλία μικρής κλίμακας και αυτό είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτά τα είδη μας ενδιαφέρουν. Ε, ε, επίσης υπάρχουν τα θέματα υγιεινής ε, για, το, για την εμπορία και τη διάθεση των αλλιευτικών προϊόντων. Έχουν δημιουργηθεί θέσεις απασχόλησης, ενισχύσαμε την καταπολέμηση της άνεργης και λαθρέας αλίας έχει σημειωθεί πρόοδο σε σχέση με την παρακολούθηση, αλλά επιδέχεται ακόμη βελτιώσει στη διαδικασία. Θέλουμε να βελτιώσουμε λοιπόν την παρακολούθηση των ελληνικών δραστηριοτήτων, την εποπτεία. Και αυτό το υπέδειξαν πολλοί συνάδελφοι στην τελευταία συνεδρίαση. Το άρθρο 10 μέσα στην έκθεση λοιπόν αναφέρεται σε αυτό και προτείνει τη σύσταση το ταχύτερο δυνατόν ενό συστήματο ε, παρακολούθηση, δορυφορική παρακολούθηση ε, του στίγματο των αλλιευτικών σκαφών που αλλιεύουν στα ύδατα του πράσινου και στην τελευταία συνεδρίαση η Επιτροπή τόνισε τη δέσμευσή τη να ε, προαγάγει την σύσταση αυτού του μηχανισμού παρακολούθηση μέσω δορυφόρου. Εγώ δηλώνω ικανοποιημένο και νομίζω ότι μιλώ εξ ονόματο και των συναδέλφων. Το νέο πρωτόκολλο συμπεριλαμβάνει και μια ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εάν υπάρχουν ε, ε, σε διεθνείς συμφωνίες τέτοιες ε, ρήτρες ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, αυτό θα μου δημιουργούσε μεγάλη έκπληξη. Νομίζω ότι είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό ε, και προβλέπεται να ανακληθεί οποιαδήποτε χρηματοδοτική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τον όρο ε, ή μάλλον αν σημειώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι σημειώθηκε παραβίαση, σοβαρή παραβίαση των αρχών της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά προβλέπονται στο άρθρο 9 της Συμφωνίας Κοτονού. υπήρξαν μεγάλα χάσματα, εντατικός ε, χάσματα απόψεων, ε, ε, εντατικό διάλογο πάνω από δύο χρόνια. Είναι υπερβολικό αυτό και ευέλπιστο ότι στο νέο πρωτόκολλο θα καλύψουμε και θα διορθώσουμε τι ατέλειε του προηγούμενου. Λοιπόν, ετησίω προβλέπονται 435.000 ευρώ σε χρηματική αποζημίωση για την πρόσβαση λοιπόν στα ύδατα, σε αυτέ τι αποκλειστικέ οικονομικέ ζώνε του πράσινου ακροτήρου. Ε, σε σχέση με το συνολικό μας προϋπολογισμό μπορεί να θεωρηθούν αυτά τα ποσά αμεληταία, αλλά έτσι 28 των αλλιευτικά και 17 ε, ε, παραγαδιάρικα και 11 δοκότρατες μπορούν να αλλιεύσουν στα ύδατα του πράσινου ακρατηρίου. Μπορούν να γίνουν κάποιες άλλες τεχνικές προσαρμογές. Θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες ε, μέσα στην ε, έκθεση. Ε, προτείνω λοιπόν ε, να δώσετε τη συγκατάθεσή σας ε, στην προσωρινή έγκριση του νέου πρωτοκόλλου και οι συνάδελφοι τόνισαν πόσο σημαντικό είναι αυτό και στα πορίσματα της συνεδρίασης της Μικτής Επιτροπής εγκρίθηκε το πολιετές πρόγραμμα και τα αντίστοιχα προγράμματα παρακολούθησης που επιβάλλει το Κοινοβούλιο. Λοιπόν, η συμμετοχή των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ιδιότητα των παρατηρητών στις συνεδριάσεις των Μικτών Επιτροπών πρέπει να κατοχυρωθεί και η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση μια πλήρη έκθεση αξιολόγηση σχετικά με την εφαρμογή του πρωτοκόλου προτού αρχίσουν νέε διαπραγματεύσει ε, για ε, μελλοντικά για ε, την έγκριση νέου πρωτοκόλλου. Ε, και το, συμβούλιο, το Κοινοβούλιο, όπως και το Συμβούλιο, πρέπει να ενημερώνεται πάρα αυτά. Αυτό προβλέπεται στη συνθήκη. Η Επιτροπή ΝΤΕΒΕ υποστηρίζει τις συστάσεις μου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας και τονίζει επίσης πόσο σημαντικό είναι να επικρατήσει η διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες για τον εντοπισμό παράνομης, ελαθρείας και ανερχή αλίας και τονίζει πόσο σημαντικό είναι να πληρούνται οι απαιτήσει πριν υποβολή αναφορών. πολέμηση επίση διαφθορά και υποβολή ετησίων εκθέσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να απευθύνονται προ το Κοινοβούλιο και προ το Συμβούλιο. Αλλά αυτά συνάδουν με τι γενικότερε διατάξει περί αποτίμηση. Δεν υπάρχουν ε, τροπολογίε επίση να υποδείξω ε, για την έκθεσή μου και ε, συστήνω να εγκρίνεται αυτή την έκθεση. Eh, Ευχαριστώ. Να περάσουμε λοιπόν τώρα στην ψηφοφορία. Υπάρχει κάποιος που δεν έχει την κάρτα του. Ωραία, έχουν όλοι την κάρτα τους. Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε η ψηφοφορία. Την έχετε βάλει ανάποδα την κάρτα σας. Εγκρίνεται λοιπόν 17 ψήφοι υπέρ, μία κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια λοιπόν κύριε Γκάλαγκερ. Εγκρίνεται η έκθεσή σας και κατά πάσα πιθανότητα θα ψηφιστεί στη δεύτερη ολομέλεια του Οκτωβρίου. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι το θέμα του προπολογισμού. Συντάκτρια της γνωμοδότησης είναι η κυρία Ρέιμερς. Έχουμε λάβει 19 τροπολογίες για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης και 30 τροπολογίες για τον προπολογισμό. Να δώσω το λόγο στην κυρία Ρέιμερ εάν θέλει να παρέμβει. Αν όχι, θα περάσουμε απευθεία στη ψηφοφορία. Κύριε Ρέιμερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες για την καλή συνεργασία. Με ενδιέφερε να στηρίξω την αηφόρα εξέλιξη της αλληλείας και να μπορέσουμε να άρουμε την ε, περικοπή των πόρων που απεφάσισε το Συμβούλιο. Δυστυχώς δεν μπορούμε πάντοτε να επιτυχάνουμε αυτό το οποίο θέλουμε και πρόκειται για την αλληλεία των ε, μικρών ακτών ε, και για τη στήριξη του τομέα κατόπιν της αυξήσεως των τιμών των καυσίμων Έχουμε λοιπόν δύο προγράμματα τώρα τα οποία στηρίζουμε διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αξιολόγησε θετικά και σας παρακαλώ να στηρίξετε αυτές τις τροπολογίες και ευχαριστώ και πάλι για την καλή συνεργασία όλους. Ευχαριστούμε και εμείς κυρία Ρέμερς. Να περάσουμε λοιπόν με τις τροπολογίες επί του προϋπολογισμού. Ψηφίζουμε την 6908 και 6924 στη γραμμή 110101 που προτείνει την αποκατάσταση του ε, σχεδίου προπολογισμού. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Στη συνέχεια, τροπολογία 6909 στη γραμμή 11.01.02.01 που πάλι προτείνει να επανέλθει ε, το ποσό στο σχέδιο του προπολογισμού. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία; Εγκρίνεται ομόφωνα. Στη συνέχεια ψηφίζουμε την 69.10 στη γραμμή 11.01.02.11 που και πάλι προτείνει να επανέλθουμε στο σχέδιο του προπολογισμού. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται ομόφωνα. Την 69-11 τώρα ψηφίζουμε στην 11 που και πάλι προτείνει να επανέλθουμε στο προσχέδιο προπολογισμού. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται 20 ψήφοι υπέρ, 2 κατά. Ψηφίζουμε τώρα την 6900 Στη γραμμή 11-01-04-03, που και πάλι προτείνει να επανέλθουμε στο προσχέδιο προπολογισμού. άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνει το 69 69-22. Στη γραμμή 11-02-01-01, παρέμβαση αλληλευτικών προϊόντων του κυρίου Φορέιρα που προτείνει αύξηση κατά 7,5 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 21 ψήφοι κατά, 1 υπέρ. Τροπολογία 69-23 στη γραμμή 11020301 για τις διεθνείς ε, συμφωνίες που παρουσίασε η ομάδα των Πρασίνων που προτείνει αύξηση σε 2 εκατομμύρια ευρώ και για τις δεσμεύσεις υποχρεώσεων και τις δεσμεύσεις πληρωμής Συγγνώμη, έκανε λάθο, Έπρεπε να ψηφίσουμε και την προηγούμενη, 6923, στη γραμμή 11020301 σχετικά με τις υπερπεριφερειακές περιοχές, ε, τις εξόχως απομακρυσμένες, ε, που προτείνει και πάλι αύξηση κατά 2 εκατομμύρια περίπου ευρώ του κ. Φεραϊρά, για την ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 19 ψήφοι κατά, 2 υπέρ και μια αποχή. Ψηφίζουμε τώρα την 6929 στην 110303 Διεθνείς Αλληλευτικές Συμφωνίες, προπαρασκευαστικές δράσεις από τους Πρασίνους, αύξηση κατά 2 εκατομμύρια σε δεσμεύσεις υποχρεώσεων και δεσμεύσεις πληρωμών. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 19 ψήφοι υπέρ, 3 κατά. Ψηφίζουμε τώρα την 6901 στη γραμμή 110611 11, Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλείας προτείνει αποκατάσταση στο προσχέδιο προπολογισμού. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 21 ψήφοι υπέρ, 1 κατά. 6902 στη γραμμή 110612 και πάλι για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλείας για το στόχο σύγκλησης που και πάλι προτείνει να επανέλθουμε στο προσχέδιο προπολογισμού άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 21 ψήφοι υπέρ, 1 κατά. 69-21 στην 11.07.01 για τη συλλογή των βασικών δεδομένων πρόταση του κυρίου Φερέιρα για αύξηση κατά 500.000 σε δεσμεύσει και 2 εκατομμύρια σε δεσμεύσει πληρωμών ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 12 ψήφοι κατά, 9 υπέρ. Ψηφίζουμε λοιπόν την ε, τροπολογία του εισηγητή στην ίδια γραμμή 6903 που προτείνει να επανέλθουμε στο προσχέδιο προπολογισμού. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας εγκρίνεται 21 ψήφι υπέρ, 1 κατά. 69-20 στη γραμμή 110702 βελτίωση των επιστημονικών γνώσεων ε, πρόταση του κ. Φερέιρα για αύξηση κατά 500.000 ε, σε δεσμεύσεις υποχρεώσεων και 1,5 εκατομμύριο σε δεσμεύσεις πληρωμών. Πέρας ψηφορίας. Απορρίπτεται 12 κατά 10 υπέρ. 6904 της εισηγήτριας, την ίδια γραμμή που ζητά να επανέλθουμε στο προσχέδιο προϋπολογισμού. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 21 ψήφοι υπέρ. 6905 στη γραμμή 110801 χρηματοοικονομική εισφορά στα κράτη-μέλη σε θέματα ελέγχου. Η συγχύτρια προτείνει να επανέλθουμε στο προσχέδιο προπολογισμού. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορίες. Εγκρίνεται ομόφωνα. 6907 στη γραμμή 11080501 για τον Οργανισμό Ελέγχου της Αλληλευτικής Κοινότητας. Η συντάκτρια της νομοδότησης προτείνει να επανέλθουμε στο προσχέδιο προπολογισμού. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται ομόφωνα. 69 28 και πάλι για τον οργανισμό κινητικού ελέγχου. Υπάρχει μια πρώτη τροπολογία των πρασίνων που προτείνει αύξηση κατά 4.200.000 επιστώσεις ε, υποχρεώσεων και 3.200 επιστώσεις πληρωμών. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 8 ψήφοι υπέρ, 13 κατά. Ψηφίζουμε λοιπόν την 6906 της συντάκτριας στην ίδια γραμμή προπολογισμού που προτείνει να επανέλθουμε στο προσχέδιο προπολογισμού. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται ομόφωνα. 69-12 τώρα νέα νομοτολογία, πιλωτικό πρόγραμμα, γραμμή 110703 της συντάκτριας. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 17 ψήφοι υπέρ, 5 κατά. Και πάλι ένα νέο πιλωτικό πρόγραμμα τώρα, 6914 για τη γραμμή 110703 του κύριου Μιλάνα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 7 υπέρ 15 κατά. Νέο πιλωτικό πρόγραμμα, τροπολογία 6915 του κυρίου Φερέιρα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 5 ψήφοι υπέρ, 17 κατά. Νέο πιλωτικό πρόγραμμα του κυρίου Φερέιρα, 69-16. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορια Απορρίπτεται. 2 ψήφοι υπέρ, 20 κατά. Νέο πιλωτικό πρόγραμμα και στην 69-17 του κυρίου Φερέιρα. Άρχεται η ψηφοφορία. απορρίπτε, συγγνώμη. Απορρίπτεται 19 ψήφοι κατά, 3 υπέρ και τελευταία τροπολογία και πάλι νεοπιλωτικό πρόγραμμα τη συντάκια 69-30, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 12 ψήφοι υπέρ, 9 κατά. Με αυτό μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία του σχεδίου γνωμοδότησης της κυρίας Ρέιμες. Όπως σας είπα και προηγουμένως, έχουμε 19 τροπολογίες και ψηφίζουμε την τροπολογία 1 της κυρίας Ρόντου, άρχη της ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Μην ανησυχείτε, εγκρίνεται. Τροπολογία 2 του κυρίου Πάξας. Άρχεται η ψηφοφορία. η ψηφοφορία; Εγκρίνεται. Η 3 είναι πανομοιότυπη, επομένως δεν την ψηφίζουμε. Τροπολογία επαριθμό 5 της συντάκτριας. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 14 ψήφοι υπέρ, 8 κατά και καταπίπτει η τροπολογία 4. Ψηφίζουμε την τροπολογία υπαριθμών 6 της κυρίας Ρόντους. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 10 ψήφοι υπέρ, 11 κατά. Η 7 του κυρίου Φερέιρα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 της εισηγήτριας λέει ο πρόεδρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 21 ψήφοι υπέρ. 10 της εισηγήτριας, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9 του κυρίου Φερέιρα ως προσθήκη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 της εισηγήτριας. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13 της κυρίας Γκρελιέ. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 9 ψήφοι υπέρ, 13 κατά. Τροπολογία 12 του κυρίου Κάντεκ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 10 ψήφοι υπέρ 12 κατά. Τροπολογία 14 του κυρίου Κάντεκ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15 του κυρίου Φερέιρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 15 ψηφικά κατά, 7 υπέρ. Τροπολογία 16 του κυρίου Φερέιρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17 του κυρίου Πάξας. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18 είναι πανομοιότυπη. Επομένως ψηφίζουμε την τροπολογία 19 της κυρίας Ρόντουστ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε τώρα το σύνολο του σχεδίου γνωμοδότησης ως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 20 ψήφοι υπέρ, μία κατά, καμία αποχή, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Ρέμερς. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και το σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης και μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης, το οποίο έχει συμπεριληφθεί κατά την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Να δώσουμε το λόγο λοιπόν στην κυρία Πατράων. Νέβη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε σχέση με αυτό το δέκατο σημείο, Θέλω πρώτα απ' όλα να προτείνω ε, για την ε, απόφαση που έγινε για την κατανομή των εκθέσεων ε, για την μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής να αναβληθεί ούτως ώστε να είναι πιο ισότιμη η κατανομή. Προτείνω από τώρα μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου που είναι η ημερομηνία της επόμενης συνεδρίας των συντονιστών, να διαβουλευτούν ε, επίσημα ή άτυπα οι συντονιστές, ούτως ώστε να βρουν μια πιο δίκαιη λύση. Κατοχυρώνοντας έτσι την ποιότητα των μελλοντικών μας εργασιών κυρίως σε σχέση με ένα τόσο σημαντικό έγγραφο, έτσι, τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Ρόντουστο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων ότι η κυρία Πατράος Νέβες έκανε αυτή την πρόταση διότι μία κοινή πολιτική αλληλείας θα πρέπει να έχει σαν τελικό στόχο να συμφωνείται με μεγάλη πλειοψηφία διότι μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να είμαστε αξιόπιστοι γι' αυτό και είμαι ευγνώμων για την κίνηση αυτή. Επίσης είμαι ευγνώμων διότι ανέφερε ότι θα πρέπει να επιζητήσουμε μία κοινή οδό να μπορούμε να συνεργαζόμαστε και στο μέλλον σε κοινό ε, και αμοιβαίο σεβασμό. Η απόφαση της 13ης Ιουλίου δεν είναι αποδεκτή για μας, γι' αυτό και πιστεύω ότι θα πρέπει να αναβληθεί ε, ο τρόπος κατανομής των εκθέσεων για να έχουμε καιρό να το συζητήσουμε μεταξύ μας, διότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να τσακωνόμαστε μέσα σε αυτή την αίθουσα. Οι ε, σοσιαλιστές, οι πράσινοι ε, και άλλες πολιτικές ομάδες δεν συμφωνούν με το τωρινό σύστημα και γι' αυτό πρέπει να μας δοθεί χρόνος να επιζητήσουμε λύσεις. Θα ήθελα να σας πω ότι θα πρέπει να επανέλθουμε στους κανόνες που έχουμε καταρτήσει, οι οποίοι αποβλέπουν στην αποφυγή διενέξεων, γι' αυτό και υπάρχουν κανόνες άλλωστε. Όταν παραβιάζονται οι κανόνες ή δεν γίνονται αποδεκτοί, υπάρχει ο κίνδυνος η συνεργασία να διακινδυνεύσει σημαντικά. Και αυτό μπορεί να μετακυλήσει και σε άλλες επιτροπές και να οδηγήσει σε ένα χάος. Οπότε κάνω μία έκκληση προς όλους να αποφύγουμε κάτι τέτοιο διότι το κοινοβούλιο μας διακρίνεται από τα εθνικά κοινοβούλια για τη δυνατότητά του να καταλήγει σε συμβιβασμό βασικές λύσεις που οδηγούν σε αποδοχή με μεγάλες πλειοψηφίες και γι' αυτό είμαι ευγνώμων στην κίνηση της κυρίας Πατράου Νέβες. Ο κύριος Γκάλαχερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ πλήρως με τη σύσταση της κυρίας Πατράου Νέβες ότι πρέπει να αναβάλουμε τη συζήτηση αυτή για να είμαστε σε θέση να λάβουμε μία απόφαση στις 19 Σεπτεμβρίου. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να έχουμε καθόλου συζήτηση και θα ήθελα να συστήσω σε εσά κυρία Πρόεδρε και στη Γραμματεία να βρει κάποια ημερομηνία για μία άτυπη συνεδρίαση των συντονιστών ή στο Στρασβούργο κατά τρόπον ώστε να έχουμε χρόνο και μία κατάλληλη αίθουση για να μπορέσουμε να διαβιλευθούμε ε, κατά τρόπον ώστε να καταλήξουμε σε μία πολιτικά ε, συνενετική πρόταση και συμφωνία. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή η πρόταση και νομίζω ότι υπάρχει και συνένεση προς το παρόν τουλάχιστον προκειμένου να προσπαθήσουμε να εξεύρουμε ένα νέο συμβιβασμό, ένα νέο τύπο που θα μας επιτρέψει να κάνουμε κατανομή. Ναι, κύριε Πατραωνέβες, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξέχασα να πω κάτι. Μίλησα για την ανάγκη να διοργανώσουμε συσκέψεις των συντονιστών μέχρι τη 19η Σεπτεμβρίου για να βρούμε μια πιο δίκαιη και ισορροπημένη λύση. Ήθελα επίσης να πω ότι το έχει προτείνει, ε, ε όπως είπε ε, και ο Ζωάο Φερέιρα προηγουμένως, ε, καλό θα ήταν να συζητηθεί αυτό το θέμα στα πλαίσια της συνεδρίασης των συντονιστών. Και άρα η πρόταση που έγινε στην αρχή της συνεδρίασης, δηλαδή η μεθοδολογία κατανομής των εκθέσεων, ε, δεν θα πρέπει να συζητηθεί εδώ, όπως είπε και ο Πάτεκο Κομπ Γκάλαχερ ε, τώρα. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε αυτήν την πιο ισορροπημένη, τη δικαιότερη λύση σε επίπεδο συντονιστών και όχι εδώ, όπως και στο παρελθόν εξάλλου. Σε αυτό το επίπεδο ε, συνεδρίασης νομίζω πρέπει να συζητηθεί το θέμα. Παρακαλώ. Ε, thank you very Ευχαριστώ εμείς από πλευρά πρασίνων διακείμεθα θετικά ε, προς τις ε, προτάσεις του ΕλΚΑ και των φιλελευθέρων να αναπενθεί δηλαδή αυτό το θέμα ή μάλλον να το πω αλλιώ, ακυρώνουμε, αν κατάλαβα καλά, την απόφαση που ελήφθη στη συνεδρία των συντονιστών και αρχίζουμε εξ αρχή ε, για να φτιάξουμε, να καταλήξουμε σε μια δικαιότερη λύση σε επίπεδο συντονιστών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε διαφανεί ως προς την κατανομή των εκθέσεων. Και επικρίνουμε τον τρόπο με τον οποίο ε, οι πολιτικές ομάδες στο παρελθόν κατέληγαν σε συμφωνία για αυτό το θέμα. Όπως ίσως ξέρουν ε, οι συνάδελφοι, στείλαμε και εμείς μια επιστολή ζητώντα μια ανοιχτή προσβάσιμη γνωμοδότηση τη νομική υπηρεσία ε, του Κοινοβουλίου σε σχέση με την κατανομή των πόντων και την πιθανή ανακατανομή αυτών των πόντων. Νομίζω ότι αυτή είναι η καρδιά του ζητήματος ε, και θα μας απασχολήσει κατά προτεραιότητα όταν θα αρχίσουμε να συζητούμε και πάλι ε, το θέμα. Αν συζητήσουμε και πάλι το σύστημα των πόντων θα διαπιστώσουμε πόσο κεντρικό είναι αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων εδώ στην Επιτροπή. Θα θέλατε εδώ με την πλήρη σύνθεση της Επιτροπής να συζητηθεί αυτό το θέμα ή να παραμείνει σε επίπεδο συντονιστών. Και κλεισμένο των θυρών, ούτως είπε. Ε, πάντως πιστεύουμε ότι είναι επιθυμητή η πλέον διαφανής διαδικασία, διότι αυτή η έκθεση είναι η πιο σημαντική που έχουμε. Έχουμε αυτή την εντολή ε, και έχουμε μια αποστολή στα μάτια των ε, ψηφοφόρων μας ε, και νομίζω ότι πρέπει με δίκαιο τρόπο να κινούμεθα. Ο κύριος Φερέιρα. Πρόεδρε, θα ήθελα να χαιρετήσω και να υποστηρίξω την ε, πρόταση επιτάπητος, δηλαδή να ξαναγίνει η συζήτηση για την κατανομή των εκθέσεων για την κοινή αλληλευτική πολιτική. Σε αυτό το πλαίσιο δεν νομίζω να υπάρξει καμία αντίρρηση σε σχέση με αυτή την πρόταση να συζητηθεί εδώ στην Επιτροπή ε, το θέμα. Ε, προφανώς η πρόταση έρχεται σε ένα πλαίσιο Εμπλοκή της κατάστασης, ε, τέλματος ε, στη συνεδρίαση ε, των συντονιστών και νομίζω ότι χρειαζόμαστε χώρο και χρόνο για να συζητήσουμε και πάλι το θέμα και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε νέα συνενετική λύση για την κατανομή των εκθέσεων. Δεν επιμένω για αυτή την πρόταση, ούτε και αντιτάσσομαι. Η συνάδελφος τώρα ε, ε πρότεινε ενδεχομένω να συζητηθεί εδώ στην, στην Επιτροπή το θέμα αυτό. Ε, δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Ε, Απλώ πρέπει να δούμε αυτό τι σημαίνει σε σχέση με την προηγούμενη απόφαση τη συνεδρία των συντονιστών. Ε, γιατί αν σήμερα λάβουμε αυτή την απόφαση, αν καταλαβαίνω ε, καλά, να μην εγκρίνουμε το σημείο 1 των πορισμάτων τη συνεδρία των συντονιστών, αυτό σημαίνει ότι δημιουργούνται οι προποθέσει τόσο σε μελλοντική συνεδρίαση των συντονιστών, να καταλήξουμε όλοι σε μια νέα λύση. Ο κύριο Γκάλεγκερ, νόμιζα ότι το πρώτο τμήμα τη συζήτηση ήταν πολύ λαριστικό και πολύ προσγειωμένο και μπορούμε ίσως να λάβουμε απόφαση να το αναβάλουμε καθώς η άλλη απόφαση που μπορούμε να λάβουμε είναι να ζητήσουμε από τη Γραμματεία να μας δώσει τη δυνατότητα να συζητήσουμε το θέμα συντονιστές και να σταματήσουμε εκεί. Αν αρχίσουμε να θέτουμε προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι η αρχή των όσων αποφασίσαμε χάνεται. Και θα ήθελα να σας ζητήσω κύριε Πρόεδρε, που δεν είμαι εγώ αυτός που θα αποφασίσει τι θα κάνουμε, να σταματήσουμε εδώ, γιατί αν συνεχίσουμε παρατέρω θα χαθεί όλη η καλή δουλειά που έχουμε κάνει και ε, θα πρέπει να προφασίσουμε να βρούμε μια συμφωνία με πολιτική συνένεση και αν οι συντονιστές είναι αυτοί που θα πρέπει να αποφασίσουμε, θα τους αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους και να έχουμε μια γενική συμφωνία. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρόντους. Ich ε, έχω μία ερώτηση κατανοήσεως προς την κυρία Πατρά Νέβε. Σωστά κατάλαβα ότι η απόφαση της 13ης Ιουλίου άρεται ότι θα ξεκινήσουμε από την αρχή και θα υπάρξει μία ε, πλήρη συζήτηση επί του θέματος. Ναι, απαντήστε, αλλά πολύ σύντομα, γιατί αλλιώ ε, ε, θα πρέπει να καθυστερήσουμε. Έχουμε πολύ κόσμο που ζητάει. Ε, θα είμαι πολύ σύντομη. τι πρότεινα. Και τέλο πάντων, ευχαριστώ για την ερώτησή σα. Εγώ πρότεινα να ανασταλεί η ψηφοφορία. Αυτό πρότεινα εγώ. Η ψηφοφορία. Δεύτερη πρόταση τώρα στο ενδιάμεσο διάστημα, δηλαδή μέχρι τη 19η Σεπτεμβρίου, θα συσκεφτούμε σε επίπεδο συντονιστών για να βρούμε μια δικαιότερη λύση. Αυτές τις δύο προτάσεις έκανα εγώ. Ο κύριος Στίβενσον. Μπορώ να σας πω ότι συμφωνώ με τον Πατ ε, Γκάλαχερ ότι μπορούμε να ε, ξεκινήσουμε εάν ε, ξαναξεκινήσουμε το θέμα για να καθορίσουμε τις προϋποθέσεις θα φάμε τη μέρα. Ας κάνουμε αυτή την ε, λογική κίνηση μίας ανεφόρων αναβολής ε, και να αφήσουμε το θέμα στους συντονιστές. Οπότε πιστεύω ότι η γραμματεία θα πρέπει να, να αναλάβει να οργανώσει μία πρώτη προκαταρκτική συνεδρίαση ίσως στο Στρασβούργο. Ούτε εγώ θέλω να πω κάτι διαφορετικό. Πιστεύω ότι είναι πολύ σοφή η πρόταση της κυρίας Πατράου Νέβε ότι ο καθένας θα πρέπει να συμβάλλει για να καταλήξουμε σε μία λογική απόφαση η οποία θα σέβεται την αντιπροσωπευτικότητα των διαφόρων πολιτικών ομάδων και τη δημοκρατία αλλά είμαι βέβαιος ότι η θα συμφωνήσουν επί του θέματος. Ευχαριστώ την κυρία Πατράο Νέβες για την τόσο λογική πρόταση. Ευχαριστώ κύριο Σαντινόρο. Δεν θα ήθελα να καθυστερήσουμε κι άλλο. Θα ήθελα να διευκρινίσω όμως το εξή. Η πρόταση που κάνει η Μαρία Πατράο Νέβες και είναι και η πρόταση της ομάδας μας και οδεύει προς την κατεύθυνση της κοινή λογικής και της αναστολής αυτού που συνέβη στις 13 Ιουλίου. Δεν θα ήθελε να περάσει το μήνυμα και σε αυτό συμφωνώ, αν κατάλαβα καλά με τα όσα είπε ο κύριος Γκάλαγκερ, ότι θα αρχίσουμε να διακυβεύουμε το θέμα της κατανομής των βαθμών και να ε, χαθεί όλα όσα ε, έχουμε επιτύχει πριν από δύο χρόνια. Υπάρχει μια απόφαση της 13ης Ιουλίου και εκεί με την κοινή λογική σε συμφωνία με τους συντονιστέ και τη γραμματεία θα μπορέσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα. Εάν όμως ξεφύγουμε προς τα μπρος, ε, να σας το διευκρινίσω εξ αρχής, δεν το δεχόμαστε. Θέλουμε απλώς να διορθώσουμε τα όσα συνέβησαν στις 13 Ιουλίου και εκεί νομίζω ότι θα μπορέσουμε όλοι να βρούμε μία καλύτερη συμφωνία. Δεν θα ήθελα να διακυβευτεί σε καμία περίπτωση αυτό που αποφασίσαμε πριν από δύο χρόνια γιατί εμείς ως πολιτική ομάδα δεν θα μπορέσουμε να το προχωρήσουμε. Ο κύριος Αντινόρο ε, έθεσε το δάκτυλο επί των ήλων γνωρίζω από κάποια πείρα που έχω συντονιστεί ότι από καιρούς καιρών κάποιες ομάδες θεωρούν ότι δεν τους αρμόζει το σύστημα των βαθμών ε, σε κάποια συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κάτι πιο σημαντικό από αυτό που συμβαίνει συνήθως. Έχουμε μία απόπειρα να ε, περικόψουμε τις πιο σημαντικές εκθέσεις που θα έχουμε στην τρέχουσα κοινοβουλευτική θητεία. Και θα ήθελα να παραπέμψουμε το θέμα στους συντονιστές ώστε να ε, ακυρωθεί η προηγούμενη απόφαση και να ξανανοίξει η συζήτηση. Και δεν είναι μόνο θέμα εμπιστοσύνη προ του συντονιστέ, αλλά οι συντονιστέ θα πρέπει να αποκαταστήσουν και την εμπιστοσύνη. Και αν το σύστημα των βαθμών δεν είναι, έχει αποτελέσματα και θα πρέπει να διαγραφεί, θα πρέπει να υπάρχει μια έκθεση προ την Επιτροπή που θα εξηγεί για ποιο λόγο γίνεται και ποιο είναι το νέο σύστημα το οποίο θα πρέπει να υιοθετηθεί προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει δικαιοσύνη νομίζω ότι έγινε μία απόπειρα για να μην υπάρχει χειραγώγηση για την κατανομή των βαθμών και των εκθέσεων. Εάν δεν λειτουργεί αποτελεσματικά το σύστημα, πέστε μας γιατί δεν λειτουργεί και διορθώστε το. Προσπαθούμε να βρούμε μια εναλλακτική συνένεση και αν δεν λειτουργεί το σύστημα των βαθμών, πέστε μας γιατί δεν λειτουργεί το σύστημα των βαθμών για αυτές τις συγκεκριμένες εκθέσεις ώστε να έχουμε μια πιο ισότιμη κατανομή, όπως ε, είπαν και οι περισσότεροι από τους προλαλήσαντες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, μου φαίνεται μένα ξεκάθαρο ότι από πλευράς κάποιων πολιτικών ομάδων αναγνωρίζουν εδώ ότι δεν ήταν ε, σωστές κάποιες από τις αποφάσεις της συνεδρίας των συντονιστών ε, και δείχνουν διαθεσιμότητα για εκ νέου συζήτηση του θέματος και χαιρετίζω αυτή του στη Βούληση. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο από τη συζήτηση. Τούτου λεχθέντος θα συμφωνήσω με την πρόταση του κυρίου Γκάλακη που επανέλαβαν και άλλοι να προσπαθήσουμε σε επίπεδο συντονιστών ήδη στο Στρασβούργο ε, να συζητήσουμε και να καταλήξουμε σε μία λύση στην επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών. Ε, τούτου λεχθέντος, αν αναγνωρίζουν αυτέ τι πολιτικέ ομάδε ότι δεν ήταν ορθή η απόφαση, ε, τότε δεν καταλαβαίνω ε, γιατί να αναβάλουμε την ψηφοφορία, την έγκριση ενό σημείου, ενώ καταλήξαμε όλοι στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν δίκαιη, δεν ήταν σωστή η απόφαση. Ε, χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό δικαιότερο σύστημα και άλλοι όροι θα διέπουν τι διαπραγματεύσει. Ε, αυτό φαίνεται να προκύπτει από τη συζήτηση. Αυτό προέκυψε από την περασμένη συνεδρία των συντονιστών. Δεν είναι πιο λογικό. Ε, δεν διευκρινίζονται έτσι περισσότερο τα πράγματα. αν υπάρχει αναγνώριση ότι δεν ήταν ορθή η απόφαση και συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να βρεθεί άλλη λύση, γιατί να αναβάλουμε λοιπόν την έγκριση αυτού του σημείου ενώ δεν είναι έγκυρο, δεν ισχύει στι μελλοντικέ διαπραγματεύσει για αυτή την απόφαση συνεδρίαση των συντονιστών από τη 13η Ιουλίου δεν είναι είναι το ενδεδειγμένο να αναβληθεί η έγκριση αυτού του σημείου λοιπόν. Καλό θα ήταν να ξανασυζητηθεί αυτό το θέμα. Μιλάω για το σημείο 1 των πορισμάτων της συνεδρίασης. Λοιπόν, αν συμφωνήσουμε ότι δεν είναι σωστή η απόφαση, ας ξεκινήσουμε εκ το μειόντος. Έτσι νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σωστό, αυτό είναι το πιο λογικό. Αφού ε, αν το αναγνωρίζουν και οι συνάδελφοι, αυτή ήταν η πρόταση, η αρχική πρόταση της κυρίας Πατραουνεύος. Αυτό είναι λογικό. Γιατί να αναβάλουμε την ψηφοφορία ενός σημείου, ενώ οι ίδιες οι πολιτικές ομάδες που κατέληξαν σε αυτή τη συμφωνία σήμερα θεωρούν ότι δεν ήταν η ορθότερη λύση. Ο κύριο Γκόρμπατσεκ για να ολοκληρώσουμε και μετά θα σας πω και εγώ την άποψή μου για τα όσα άκουσα από του περισσότερους εξημών. Κύριε Γκόρμπατσεκ από την πλευρά μου <clears throat> θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια. Ακούσαμε ορισμένες προτάσεις και την επόμενη εβδομάδα μπορούμε να έχουμε μία περαιτέρω συνεδρίαση και θα πρέπει να φροντίσουμε η απόφαση η οποία θα ληφθεί από τους συντονιστές να μπορέσει να αντικατοπτρίζει και την ε, άποψη της πλειοψηφίας της ομάδος. Ωραία, λαμβάνοντα υπόψη την άποψη τη πλειοψηφία, νομίζω ότι θα πρέπει να αναβάλουμε οποιαδήποτε απόφαση, τουλάχιστον για σήμερα. Θα οργανώσουμε στο Στρασβούργο μία συνεδρίαση, άτυπη συνεδρίαση των συντονιστών, με στόχο να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε ένα νέο συμβιβασμό, σε μία συνένεση, σε μία νέα συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων, ώστε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θα σας ανακοινώσουμε πότε μπορούμε να έχουμε αίθουσα με διερμηνία, μία μέρα η οποία θα ευνοεί τους πάντες και θα κάνουμε μία απόπειρα να κάνουμε τη συνεδρία σε αυτή στην επόμενη Ολομέλεια του Στρασβούργου. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε. Ευχαριστώ τις πολιτικές ομάδες ε, που επέδειξαν διάθεση να καταλήξουμε σε μια νέα συνένεση που θα είναι ευρύτερη και θα περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερες πολιτικές ομάδες. Και λοιπόν αυτό θα κάνουμε που σας ανακοίνωσα. Ολοκληρώνεται λοιπόν το συγκεκριμένο σημείο στην ημερήσια διάταξη και περνάμε τώρα στη Συμφωνία για το Μαρόκο. Έχουμε δύο σημεία. Έχουμε καταρχάς το σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης που αφορά το Μαρόκο. Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Μαρόκου σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωση για τα γεωργικά προϊόντα και τα αλλιευτικά προϊόντα. Η συγητή, συντάκτη συγγνώμη τη γνωμοδότηση είναι ο κύριο Ρωμέβα Ιρουέδα. Ο κύριο Ρωμέβα μα έχει ήδη παρουσιάσει κάποια πράγματα, έγινε μια συζήτηση, παρουσιάστηκε και η γνωμοδότηση της ε, νομικής υπηρεσίας και τώρα ο κύριος Ιρουέδα θα μας παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησης που έχει εκπονήσει. Να σας δώσω λοιπόν το λόγο για να μας παρουσιάσετε το σχέδιό σας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών ε, ήρθαν σε επαφή μαζί μας, το προσωπικό της γραμματείας καταρχάς, αλλά και η ε, υπηρεσία διερμηνίας και μετάφρασης, η οποία μας βοήθησε να έχουμε έτοιμα τα κείμενα σήμερα. Παρά τι καλοκαιρινέ διακοπέ, μπορέσαμε να τα καταφέρουμε. Υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία έπρεπε να διορθωθούν αυτέ τι μέρε και τα καταφέραμε και επομένω, ελπίζω να έχετε όλοι την ε, γνωμοδότηση στη γλώσσα σα επικαιροποιημένη. Όπως γνωρίζετε, πρόκειται για γνωμοδότηση. Μία γνωμοδότηση για μία έκθεση για την οποία είναι αρμόδια επί της ουσίας η ΙΝΤΑ και έχουμε τις επιπτώσεις ε, για τα αλληλευτικά προϊόντα και την αλληλευτική διάσταση. Έχουμε τη συμφωνία με το Μαρόκο, συμφωνία σύνδεσης, ε, η οποία αναθεωρείται επί του παρόντος και υπάρχουν κάποιες πτυχές οι οποίες ε, είναι κοινέ κατά την άποψη της Επιτροπής μας και με τα όσα λέει ο βασικός ε, συντάκτης της, ε, της ε, έκθεσης, ο Ζωζέ Μποβέ. Υπάρχουν κάποια σημεία που σας απασχολούν και ήθελα να τα θίξω στη γνωμοδότηση αυτή. Καταρχάς, να υπενθυμίσω ότι η συμφωνία αυτή θα επιτρέψει την απελευθέρωση των εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 55% και ταυτόχρονα τις εισαγωγές από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Μαρόκο συγγνώμη, από πλευρά Μαρόκου διορθώνει ο μιλητή, θα είναι κατά 45%. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Αλλά αυτό που μα ενδιαφέρει εδώ δεν είναι τόσο η ποσότητα όσο η ουσία. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι εισαγωγές αυτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε προϊόντα τα οποία προέρχονται από το Μαρόκο με ανοιχτά όμως ζητήματα όπως για παράδειγμα ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι έλεγχοι και πώς ε, ε τηρούνται οι προθεσμίες και οι ποσοστώσεις ε, και οι δεσμολογικές ε, πτυχές Ακούσαμε ε, εμπειρογνώμονες του κλάδου και εκπροσώπους του κλάδου σε αρκετές περιπτώσεις και υπάρχουν και πάρα πολλές αμφιβολίες διότι δεν ξέρουμε κατά πόσον οι ίδιες προϋποθέσεις που ζητείται να τηρούνται από τους ε, υπευθύνους του τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τηρούνται και από το Μαρόκο. Αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο το οποίο θεωρούμε ότι είναι πολύ ουσιαστικό και θα πρέπει να το επισημάνουμε. Δεν πρόκειται για εντύπωση, αλλά υπάρχουν μία σειρά από ανησυχίες οι οποίες μας ήρθαν από διάφορες οργανώσεις που ε, ενδιαφέρονται άμεσα ή έμεσα για το ζήτημα. Δεύτερο στοιχείο, το οποίο έχει σχέση περισσότερο με την Επιτροπή μας. Αρκετές εκθέσεις, τις οποίες ε, διευκρινίζεται σαφώς η κακή ή πολύ κακή κατάσταση των αποθεμάτων ε, στα ύδατα του Μαρόκου. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια σχετική έκθεση και θα έπρεπε και αυτό σας το λέω ιδιαιτέρως ότι θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί όταν θέλουμε να εγκρίνουμε νέους κανόνες για την εισαγωγή νέων προϊόντων τα οποία επιμένω ότι θα μπορούσαν να προέρχονται από αποθέματα τα οποία είναι πλήρως εξαντλημένα ή εξαντλούνται, ε, θα εξαντληθούν πολύ σύντομα. Επίσης, μας ενδιαφέρουν οι γεωγραφικές ενδείξεις. Είναι κάτι το οποίο είναι όλο ένα και πιο σημαντικό και το έχουμε επαναλάβει πολλές φορές εδώ στο Κοινοβούλιο. Ε, οι καταναλωτές και οι καταναλώτριες θα πρέπει να γνωρίζουν από πού προέρχονται τα προϊόντα που καταναλώνουν. Και επομένω, οι γεωγραφικές πληροφορίες και για τα προϊόντα αυτά είναι ζωτική σημασία. Υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες ε, διότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να καθορίσουμε σαφώς τη γεωγραφική προέλευση κάποιων προϊόντων. Ορισμένες φορές αναφέρεται απλώ το Μαρόκο ή και λαμβάνονται και ευρωπαϊκές ετικέτες ακόμα και αν δεν προέρχεται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα προϊόν αλλά από άλλες περιοχές και πρόκειται για μια πρακτική που δεν είναι απαραίτητο παράνομη αλλά μπορεί να δημιουργήσει κάποιες δυσκολίες από, για τους καταναλωτές και για τα συγκεκριμένα προϊόντα. Ένα τελευταίο στοιχείο το οποίο δεν είναι ίσονο σημασία, είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα το οποίο έχει σχέση και με αρκετές συζητήσει που κάνουμε και νομίζω ότι είναι και το πιο διαφιλονικούμενο ζήτημα. Είναι το ζήτημα που έχουμε αναφέρει επανειλημμένως της Δυτικής Σαχάρας. Εδώ υπάρχουν στοιχεία τα οποία ταυτίζονται και με ένα άλλο παράλληλα ζήτημα που συζητάμε, είναι η Αλευτική Συμφωνία με το Μαρόκο, την οποία θα δούμε στη συνέχεια. Και υπάρχει ένα ουσιαστικό πρόβλημα, ένα βασικό πρόβλημα, το οποίο δεν θα πρέπει να λησμονούμε. Κάθε άλλο θα πρέπει να προσπαθούμε να βρούμε μία λύση, διότι κάθε φορά τίθεται το, το ίδιο ζήτημα και κάθε φορά είναι όλο και πιο περίπλοκο να ξεύρουμε μία λύση επί του ζητήματος αυτού. Eh, Όταν λοιπόν ζητάμε από το Κοινοβούλιο να μας πει εάν θα συμπεριληφθεί η Δυτική Σαχάρα στο πλαίσιο εφαρμογής του Συμφωνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας απάντησε σαφώς ότι εφόσον οι εξαγωγές ε, έχουν συγκεκριμένες ε, προτιμήσεις, εμπορικές προτιμήσεις, τότε θα γίνονται ε, δεκτά. Η συγκεκριμένη πρόταση ήταν στο μέτρο που εξαγωγή προϊόντων από τη Δυτική Σαχάρα ήδη υποφελούνται εμπορικών προτιμήσεων. Θα πρέπει όμω να δούμε και τι επιθυμεί ο πληθυσμό τη Δυτική Σαχάρα. Γι' αυτό λοιπόν επαναλάβαμε την ερώτησή μα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ρωτήσαμε κατά πόσον ήρθαν σε επαφή με τον πληθυσμό τη Δυτική Σαχάρας και του νόμιμου εκπροσώπου για να μάθουμε ποιε είναι οι επιθυμίε του. Και η απάντηση που λάβαμε είναι ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο και έτσι διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε καμία ενημέρωση. Καταρχάς για το πώς εποφελούνται από τις συμφωνίες αυτές οι κάτοικοι της Δυτικής Σαχάρας και δεύτερον πώς ε, α... πλήττεται ο τοπικός πληθυσμός ή εποφελείται και επειδή δεν μας έδωσε επισήμως απάντηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εγώ προσπάθησα να έρθω σε επαφή με τους ενδιαφερομένους για να μάθω την άποψή τους. Θεωρώ ότι είναι καθήκον μου άλλωστε να το κάνω και έτσι είχαμε και την άποψη των ενδιαφερομένων. Πρόκειται για το κείμενο το οποίο έχετε στη γνωμοδότηση. Το έχω γράψει λέξη προς λέξη για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποιες είναι οι προτάσεις και οι συγκεκριμένες σκέψεις που προκύπτουν από την ε, ε, πλευρά αυτή. Και σε γενικέ γραμμέ αυτέ είναι οι τέσσερι πτυχέ που με ανησυχούν ε, στη γνωμοδότηση. Πρόκειται για μια σειρά από ανησυχίε, αμφιβολίε, από ερωτήσει που δεν έχουν λάβει απάντηση και αυτό με υποχρεώνει να ζητήσω από πλευράς ε, της Επιτροπής μας η γνωμοδότηση για την αναθεώρηση της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου με το Μαρόκο να ζητήσει απόρριψη ή επανεξέταση. Υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις δεν ε, έγιναν πολλά από τα θέματα τα οποία θα ε, πίστευα ότι θα έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί και γι' αυτό πιστεύω ότι η Επιτροπή μας δεν θα ήθελε να προχωρήσουμε, τουλάχιστον όχι από αυτού τους όρους με την ε, πρόταση αυτή. Και αυτή λοιπόν είναι και η τελική μου πρόταση όπως θα διαβάσετε στο κείμενό σας, το Κοινοβούλιο να αρνηθεί αυτή την σύμφωνη γνώμη γιατί δεν θεωρούμε ότι είναι σωστά αυτά τα οποία προκύπτουν από την αναθεώρηση τη συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου. Ε, είμαι στη διάθεσή σα για να ακούσω προτάσεις, ε, για να δούμε και πώς ε, θα έχει η τελική θέση τη επιτροπή μα. Επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για μια γνωμοδότηση, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει και μια ταύτιση απόψεων με τη βασική συζήτηση που γίνεται στην αρμόδια επί Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Ανδρέα Μπαρέα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση, μια γνωμοδότηση ε, η οποία έχει μια επιτυσσουσία αρμόδια επιτροπή και έχουμε μια πολύ σημαντική πολιτική βάση, μια πολύ σημαντική και συναισθηματική βάση και λίγο πολύ αυτή η συμφωνία ε, συζητιέται. Μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων και 22 Νοεμβρίου θα παρουσιαστεί η έκθεση. Για το Μαρόκο και για τις συμφωνίες του, είτε τις αλλιευτικές είτε τις εμπορικές συμφωνίες, έχουμε συζητήσει επανειλημμένως ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα και ε, έχουμε πάντα το ίδιο πρόβλημα που έχουμε συνήθως, το εδαφικό πρόβλημα. Εγώ επανειλημμένως εδώ στην Επιτροπή έχω πει ότι αν αφήσουμε στην άκρη το εδαφικό στοιχείο, το οποίο είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα μπορεί με να μας αφορά προσωπικώς, αλλά δεν είναι αρμοδιότητα αυτής της Επιτροπής, η συμφωνία αυτή σε γενικές γραμμές, η εμπορική συμφωνία για την... Ε, Επιτροπή και τη συμφωνία αυτή αυτή ήταν ικανοποιητική, διότι υπάρχει εξαγωγή από πλευράς Μαρόκου και ε, εισαγωγή από πλευράς Μαρόκου ε, από Ευρωπαϊκή Ένωση και το ίδιο ύφελος έχουμε και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και εξαγωγές και εισαγωγές υπήρξαν επικρίσεις. Στην Ισπανία υπήρξαν επικρίσεις από τις γεωργικές ε, ενώσεις, ε, πολύ σημαντικές επικρίσεις για τις ε, αύξηση των ελέγχων και ούτε καθεξής, αλλά έχουμε μια νέα συμφωνία και αυτή η νέα συμφωνία θα μπορούσε να φροντίσει να ρυθμιστεί αυστηρότερα το ζήτημα αυτό και να υπάρχει περισσότερος έλεγχος για τους υγειονομικούς ελέγχους. Όσον αφορά τώρα τα ωφέλη, Πράγματι υπάρχουν ε, μεγάλες δυσκολίες και δεν ξέρουμε κατά πόσον επωφελείται η Δυτική Σαχάρα από τους τομείς ε, αυτούς, από τα ωφέλη αυτά. Αλλά ε, θα πρέπει να κάνουμε ελέγχους για να ξέρουμε για τα γεωργικά προϊόντα τουλάχιστον πού παράγονται. Στην έκθεση που ε, ετοιμάζει η Επιτροπή ΙΝΤΑ βρισκόμαστε ακόμα σε προκαταρκτικό στάδιο. Νομίζω όμως ότι είναι νωρίς ακόμα και δεν μπορούμε να πούμε ότι θα πρέπει να απορρίψουμε τη συγκεκριμένη πρόταση. Θα πρέπει να δούμε και τι εργασίες θα κάνει η αρμόδια επί της Επιτροπή και να προσπαθήσουμε να έχουμε μια ισορροπία και θα προσπαθήσουμε να μην έχουμε μεγάλες διαφορές με άλλες συμφωνίες. Εάν υπάρχει και άλλη συμφωνία ε, άλλες συμφωνίες που έχουν οι ίδιες ε, πτυχές γιατί να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά εδώ στη συμφωνία με το Μαρόκο. Ε, θα πρέπει να δούμε τι ε, συμφωνία γίνεται βάσει των συμφερόντων της Επιτροπής μας και όχι των προσωπικών μας απόψεων. Ευχαριστώ κυρία madam. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι ανάμεσα ε, στα φρέσκα ψάρια και τα φρέσκα ψάρια σε κονσέρβα υπάρχει κάποια διαφορά. Ε, αυτά τα προϊόντα αντιστοιχούν στο 11% των συνολικών εσόδων από τις εξαγωγές για το Μαρόκο, παραπάνω δηλαδή από ότι τα γεωργικά προϊόντα και το 70% των ψαριών αυτών προορίζονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι δικό μας ε, θέμα. Ε, βάσει αυτη της αλλιευτικής συμφωνίας γνωρίζουμε ότι ε, δεν είναι καλή η κατάσταση των αλλιευμάτων. Ξέρουμε όλα αυτά περί Δυτικής Σαχάρας κτλ. Σε προηγούμενη συνεδρίαση είχα σχολιάσει αυτό το θέμα, δηλαδή η, ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε σχέση με προϊόντα που έρχονται από κατεχόμενα, προέρχονται από κατεχόμενα εδάφη. Ε, η Γάζα, Δυτική Όχθη, τα υψώματα του Γκολάν, ε, Ανατολική Ιερουσαλήμ, ε, στο Ισραήλ. Αν θεωρούνται δηλαδή Ισραηλινά προϊόντα και ως εκ τούτου εντάσσονται σε Συμφωνία Ελευθερού Εμπορίου με το Ισραήλ ή όχι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεώρησε ότι αυτά τα υψώματα Γκολάνε, Δυτική Όχθη κτλ. δεν μπορούν να θεωρηθούν ως τμήμα των εδαφών του Ισραήλ. Ε, αυτό προκύπτει από το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας ε, του ΟΗΕ και αυτό απηχείται επίσης με μια ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή ε, της Εμπορικής Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ που δημοσιεύθηκε το 1988. Δυνάμει αυτή τη συμφωνία, η ζώνη ελευθέρου εμπορίου που καλύπτεται από τη συμφωνία δεν καλύπτει αυτά τα κατεχόμενα εδάφη. Η Λίδια Άστον έδωσε μία απάντηση σχετικά με το αν η Δυτική Σαχάρα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο Μαρόκο ή όχι και άρα να καλυφθεί από αυτή τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ Μαρόκο. Αυτό δεν προκύπτει με σαφήνεια. Η νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέφερε ότι τα εδάφη της Δυτικής Σαχάρας στην άμυ του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να θεωρηθούν ότι αποτελούν στο κομμάτι ε, το, της επικράτειας του Βασιλείου του Μαρόκου. Άρα έλλειψη ε, σαφήνειας από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θεωρεί ότι διοικείται ε, νομίμως και θεμητά ε, η Δυτική Σαχαρά από το Μαρόκο. Αν δεν το πιστεύουμε αυτό θα έπρεπε να έχουμε αντίστοιχη δήλωση για τη Δυτική Σαχάρα όπως εκείνη που λάβαμε για την ε, λωρίδα της Γάρας στα υψώματα του Γκολάν και τη Δυτική Όχθη. Θα ήθελα λοιπόν να στραφώ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, εξηγήστε μας ε, τη διαφορά στην μεταχείριση ως προς αυτές τις δύο ε, προαναφερθείς εμπορικές συμφωνίες. Αυτό που βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι συζητούμε τώρα αυτό το θέμα μετά το καλοκαίρι, μετά την Αραβική Άνοιξη και με όλες τις λαϊκές εξεγέρσεις που έγιναν στη Βόρεια Αφρική και εμείς ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι οι επιθυμίες των αυτοχθών δεν συμπίπτουν όποια έκπληξη ε, με τις επιθυμίες και τις ανάγκες ε, των ε, όσων διοικούν αυτές τις χώρες τις δικτατορίες. Οπότε οι επιθυμίες των, των λαών, των φυλών της Δυτικής Σαχάρας έχουν ζωτική σημασία τώρα και δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή είναι να δείξει ότι είμαστε στο, ε, στην πρώτη γραμμή στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σεβόμαστε τα δικαιώματα όχι μόνο αυτών που είναι στη Βόρεια Αφρική αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά τώρα αυτό μας απασχολεί. Η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με το Μαρόκο ε, και τη Δυτική Σαχάρα και δεν ξέρουμε αν υποφελούνται ε, οι αυτόχθονε φυλέ από αυτή την ε, συμφωνία. Έχουμε μάλιστα αντίστοιχες ε, ενδείξεις ότι αυτό δεν συνάδει με τις επιθυμίες τους. Εξηγήστε μου σας παρακαλώ τη διαφορά μεταχείρισης ανάμεσα στα κατεχόμενα της Δυτικής Αχάρης και τα κατεχόμενα από το Ισραήλ. Θα με βοηθούσατε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ τον συντάκτη της γνωμοδότησης για την άποψή του. Έθεσε μία σειρά από ανησυχίες, ε, καθόλου λογικές. Θα πρέπει να δούμε τη γνωμοδότηση στα πλαίσια της Επιτροπής Αλίας Υπάρχει μια συμφωνία Ρομέντ από το 2000 ε, και υπάρχει και το άρθρο 16 που λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία εμπορικής ελευθέρωσης των προϊόντων. Ε, μέχρι τούδε προέκυψε ότι υπάρχει ε, μεγάλο εμπορικό συμφέρον μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάγει στο Μαρόκο το διπλάσιο αυτών που εισάγει και είναι προφανές ότι είμαστε υπέρ της εντατικοποίησης των εμπορικών σχέσεων με το Μαρόκο και αναφέρομαι τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο Μαρόκο. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να ε, δώσουμε νέα κίνηση στην οικονομία εκατέρωθεν και να υπάρχει ένας δημοκρατικός χώρος, χώρος ευημερία στη Βόρεια Αφρική καθώς επίσης και να συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη της οικονομίας ε, στο Μαρόκο και τη μείωση της ένδυας. Θεωρώ ότι κάποια από τα θέματα τα οποία αναφέρθησαν έχουν επιληθεί στο κείμενο της συμφωνίας. Κάποια άλλα είναι θέματα γενικού χαρακτήρα. Ε, τους ελέγχους, για παράδειγμα, που αναφέρεται ε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ή στους ελέγχους στο Μαρόκο, αλλά μας ενδιαφέρει και το σύνολο των εξαγωγών και εισαγωγών που μπορεί να γίνει και θα πρέπει να το σκεφτούμε λίγο πιο γενικά και να μην υπάρχει μόνο κάτι συγκεκριμένο για μια συγκεκριμένη συμφωνία. Στη συμφωνία έχουμε μέτρα διαφύλαξης, υπάρχουν και κάποια υγειονομικά και φυτοϊγειονομικά μέτρα. Στο άρθρο 7 αναφέρονται και το πλαίσιο επίλυσης. Είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά ε, και τα όσα έχουμε για το εμπόριο εν γέννη. Υπάρχουν και συμφωνίες σε υπουργικό επίπεδο για να προχωρήσουμε όλες αυτές τις πτυχές, περισσότερες γεωγραφικές ενδείξεις. Ε, στο άρθρο 8 του πρωτοκόλου αναφέρεται και ότι τρεις μήνες ε, μετά από την έναρξη ισχύω του πρωτοκόλου θα ξεκινήσει και μια συζήτηση για τις γεωγραφικές ενδείξεις με στόχο να καταλήξουμε σε συμφωνία εντός ενός έτους και όσον αφορά το θέμα της δυτική ε, Σαχάρα, υπάρχει και μια επιστολή της, επί, ε, της, εκπροσώπου Άστον που αναφέρεται στην περίπτωση της Δυτικής Σαχάρας θα υπάρξει ένας μηχανισμός για την ε, παρακολούθηση της εφαρμογής της συγκεκριμένη συμφωνίας. Η κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα είναι μία περιοχή η οποία είναι διαφιλονικούμενη και πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε τα όλα αυτά τα θέματα, θα πρέπει να αξιολογήσουμε και τις οικονομικές ε, συνέπειες που μπορούμε να έχουμε και δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε προσκόμματα τα οποία ε, θα είναι κατά των συμφερόντων της ε, Επιτροπής μας. Θα πρέπει να δούμε ε, τι είναι το καλύτερο για την Επιτροπή μας και να μην σταθούμε μόνο στα προβλήματα της Δυτικής Σαχάρας. Ο κύριος Φερέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω για την παρουσίαση της έκθεσης και να τονίσω ε, την πληρότητα της έκθεσης αυτής. επενώ τον εισηγητή, ε, διότι μας παρουσίασε όχι μόνο την οργάνωση του κλάδου εδώ στην Ευρώπη, αλλά ε, υπερβαίνει ε, ένα συγχώρητο, μια συγχώρητη παράληψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τους εκπροσώπους των Σαχράουι στη διεθνή σκηνή. Νομίζω πρέπει να το τονίσουμε αυτό γιατί προσδίδει μια αρετή στην έκθεση που να αξιέπινη. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι άλλο. Ε, πρόκειται για αλλιευτική συμφωνία, το οποίο είναι και πάρα πολύ ε, διαφορετικό σε σχέση με άλλες συμφωνίες. Πρόκειται για μια συμφωνία απελευθέρωσης ε, του εμπορίου που συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων τα αλλιευτικά προϊόντα. Θα ήθελα εδώ να θυμίσω μια συζήτηση που είχαμε εδώ στην Επιτροπή μας όταν ο συνάδελφος Καντέκα συνέτασε την έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις απελευθέρωσης ε, του διεθνούς εμπορίου ε, στον τομέα ε, των αλλιευμάτων των προϊόντων αλλίας. Σε εκείνη τη συζήτηση... Α, και να πω ότι έτυχε ευρεία αποδοχή η έκθεση στην Επιτροπή μα. Κατέδειξε λοιπόν ε, τι ε, παράπλευρε αρνητικέ επιδράσει απελευθέρωση του διεθνού εμπορίου στον τομέα τη ε, τότε είχαμε σωστά υποδείξει ε, αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε λοιπόν ε, εδώ να συμβεί ε, το αντίθετο γιατί έχουν εκφραστεί ανησυχίες από τον κλάδο και ακούσαμε και τις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας και από τους συναδέλφους σχετικά με την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα. Πέρα από το θέμα της ε, Δυτικής ε, Σαχαράς, όχι ότι δεν είναι σημαντικό το θέμα, αναφερθήκαμε και στα ε, πρότυπα υγιεινής. Αναφέρει ο εισηγητής αυτό το σημείο της μη τήρησης των κανόνων υγιεινής δεν υπάρχουν σχετικές διατάξεις ούτε και προστασίας του περιβάλλοντος δεν υπάρχουν πρότυπα στον τομέα της εργασίας της κοινωνικής ασφάλειας δεν πρέπει να ξεχνάμε, δεν μπορούμε ε, να ξεχνούμε πέρα από τα θέματα υγιεινής την ε, ε, πασιφανή έλλειψη κοινωνικών προτύπων, προτύπων κοινωνικής ασφάλισης που είναι όμως ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της συμφωνίας. Προφανώς δεν ικανοποιείται κατά πρότυπα που ισχύουν στο Μαρόκο. Τώρα το θέμα της Δυτικής Σαχάρας. Πρόσπαθη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάλι και λυπούμε γι' αυτό ε, η Πούλα προσπαθεί να εισαγάγει αυτή τη συμφωνία στα εδάφη της Δυτικής Σαχάρας αγνοώντας ε, το πρόβλημα. Ε, και ανεξάρτητα από αυτά που ακούσαμε από τους συναδέλφους, γιατί αυτό δεν σχετίζεται μόνο με αυτή τη συμφωνία, αλλά είναι ευρύτερο και σχετίζεται, όπως είπε ο συνάδελφος Σάντες και Μπαρέια, σχετίζεται λοιπόν αυτό το θέμα και με τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μαρόκου γενικότερα. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι πρέπει σε κάποιο άλλο φόρουμ να συζητηθεί αυτό το θέμα και να εγκρίνουμε ακέραιη την έκθεση. Ε, εντάξει, η έκθεση καλύπτει και άλλα σημεία, αλλά και αυτό ε, και η λύση που θα βρεθεί θα επηρεάσει και αυτή τη συμφωνία. Δεν μπορούμε να αγνοούμε ε, τη συμφωνία, να εθελοτυφλούμε και όπω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή πουλά, το ξαναλέω, ε, να εισαγάγει αυτή τη συμφωνία στη Δυτική Σαχάρα για να υποφεληθούμε από τα προϊόντα τη. Μα είναι θέμα διεθνού δικαίου. Ε, υπάρχει θέμα και η νομική υπηρεσία είχε εκφράσει μια, σε μια γνωμοδότησή τη την ανησυχία τη για αυτά τα θέματα διεθνού δικαίου. Λοιπόν, αντιμέτωποι με αυτά τα θέματα, τονίζω και πάλι, δεν είναι μόνο το θέμα της Δυτική Σαχάρα που έχει καθοριστική σημασία, αλλά και για αυτό το θέμα, αλλά και για άλλα. Κρίνω πως ε, η έκθεση ε, θα πρέπει να προτείνει να απορριφθεί αυτή η πρόταση συμφωνίας απελευθέρωσης του εμπορίου στη μορφή που έχει τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι προχωράμε αργά και σκέφτομαι ότι όντως ένα πρωτόκολλο πρέπει να επιτρέψει ένα πολιτικό πλαίσιο για την εφαρμογή αυτής της αλλιευτικής συμφωνίας η οποία δεν λύνει τα προβλήματα των εδαφικών εντάσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή αλλά όλοι γνωρίζουν ότι αν δεν υπάρξει μία τελική λύση σχετικά με την αυτονομία και τη δυνατότητα να ισχύσει σαν ανεξάρτητο έδαφος με ε, πολιτική ε, διεθνή οντότητα ε, υπάρχει μια έλλειψη η οποία δεν θα λυθεί από την αλλιευτική συμφωνία. Μέσα λοιπόν στην παρούσα κατάσταση πιστεύω ότι προς το λαό της Σαχάρας και του Μαρόκου θα πρέπει να διευκρινίσουμε την κατάσταση. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την κατάσταση της Παλαιστίνης ε, με αυτήν ε, της Σαχάρας, με την Αλγερία και το Μαρόκο γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι μόνο αυτοί οι συνομιλητές οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτό το χώρο της Βορείου Αφρικής και γι' αυτό πιστεύω ότι η Επιτροπή μας δεν θα λύσει το ουσιαστικό πολιτικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει αλλά απλώς πρέπει να επαληθεύσει ότι ε, υπάρχει μία συμφωνία η οποία εφαρμόζεται σύμφωνα με τις διαπραγματεύσεις. Μία εμπορική συμφωνία πρέπει να εξετάζεται από την οπτική γωνία της δικαιοσύνης ε, εμπορικά και από τις δύο πλευρές για να υπάρχει λοιπόν μία σύγκληση μεταξύ ε, των θέσεων της Επιτροπής Ίντα και αλλιώς θα ήθελα να εφαρμόσουμε την ε, ε, ρήτρα διαφυγής ε, για να τονίσουμε τα ωφέλη που μπορεί να αποκομίσει ο λαός της Σαχάρας και πιστεύω ότι αυτή η συνέπεια είναι σημαντική. Όσον αφορά το πολιτικό περιβάλλον, ξέρω ότι το ανέφερε η κυρία Άστον, δεν πρέπει να πω ότι, δεν μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένη με την αντιμετώπιση αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι μαζεύουμε τα σπασμένα όπως το είπε και ο εισηγητής και θα πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία. Δεν θα μπορέσουμε με μια κίνηση να λύσουμε όλα τα προβλήματα και δεν νομίζω ότι η απόρριψη της σωστής πολιτικής μπορεί να ισχύσει. Πρέπει να προχωρήσουμε με διαφάνεια, με δυνατότητες εγγυήσεων από όλε τι πλευρές, διότι σε αυτό το ρευστό πολιτικό κλίμα χρειάζεται υπευθυνότητα εκ μέρους των αρχών του Μαρόκου, νεαρούς των συνομιλητών της Σαχάρας, των Ευρωπαίων και όπως ε, είπε προηγουμένως και ο συνάδελφός μου, καλό θα ήταν να μπορέσουμε να προχωρήσουμε θετικά στα πλαίσια αυτά και στηρίζω την ε, κίνηση την οποία στήριξαν πολλοί από τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος άλλος? Ωραία, να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη Γενική Διεύθυνση Trade την Κοινωνική Διεύθυνση Εμπορίου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, είμαι από την ε, ε, υπάρχει βέβαια η υπηρεσία εξωτερικής ε, δράσης που θα μπορέσει επίσης να σχολιάσει το θέμα αυτό αλλά σαν εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου πρέπει να σχολιάσω τρία σημεία σε αυτή τη συμφωνία. Όταν διάβασα αυτό το σχέδιο ψηφίσματος ε, αναρωτήθηκα διότι θυμάμαι ότι πέρυσι το Δεκέμβριο έγινε μία συζήτηση επί της ουσίας αυτής της συμφωνίας και ουσιαστικά υπήρχε μία θετική αξιολόγηση στην Επιτροπή αυτή από όσου έλαβαν το λόγο και οι οποίοι χαιρέτησαν τη συμφωνία αυτή εκτός από τα σχόλια σχετικά με τα ιδεαφικά θέματα. Ε, βλέπω όμως τώρα ότι η μόνη εξήγηση την οποία μπορώ να δώσω είναι ότι υπάρχει μία σύγχυση και συνδέει κανείς υπερβολικά την αλληλεία με την γεωργία στο σχέδιο ψηφίσματος γνωμοδότησης ε, ε, του εισηγητή διότι ζητείται μία απελευθέρωση και αυτό είναι ένα λάθος ουσιαστικό ε, διότι αν θυμάστε το 1996 η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ήδη απελευθερώσει μονομερός 100% το θέμα έναντι του Μαρόκο και ίσχυσε αυτό από το 2000 όλα λοιπόν τα προϊόντα του Μαρόκο ε, εισάγονται εις ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αγορές της χωρίς πότους σωστό Οπότε πρέπει να υπάρξει ε, ένας ισοσκελισμός. Γι' αυτό και ζητήσαμε ορισμένες υποχωρήσεις για προϊόντα από την Ευρώπη που οδεύουν προς τις μαροκινές αγορές. Ε, ε, αυτή είναι η κατάσταση με τους μαροκινούς ομολόγους μας και όπως σας είχα πει και πέρυσι το Δεκέμβριο πρόκειται για ουσιαστικές υποχωρήσεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και εμείς θα εξάγουμε στο Μαρόκο για την επόμενη πέντα ετία ότι ε, θα ανταποκρίνεται σε 91% των μαροκινών προϊόντων που θα εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς δασμούς και στο θέμα αυτό η εφαρμογή εφαρμογή των ποσοστώσεων, δασμολογικών ποσοστώσεων δεν έχει κανένα νόημα διότι κάποια ημέρα θα υπάρξει μία πλήρης απελευθέρωση και ούτως ή άλλως από το 2000 τα μαροκινά προϊόντα εισέρχονται στην Ευρώπη χωρίς ποσοστώσεις και χωρίς καμία παρέμβαση αγοράς. Ε, θεωρούμε λοιπόν ότι με αυτή την απελευθέρωση απλούστατα θα οξύνουμε την ισχύ Σα κατάσταση των ε, μειωμένων αποθεμάτων ε, ψαριών εις τα μαροκινά ύδατα και οι συζητήσεις οι οποίες γίνονται δεν θα αλλάξουν σημαντικά ε, το σκηνικό αυτό. Επίσης, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η υπάρχουν ε, ενδείξεις για ορισμένα μέσα ε, που άπτονται παραδείγματος χάρη ε, συγκεκριμένων προϊόντων όπως η παρμεζάνα, η μουστάρδα της Dijon που αναφέρονται στην ονομασία προελεύσεως. Αν υπάρχει λοιπόν σήμανση προελεύσεως για τον καταναλωτή θα πρέπει ε, να μπορεί κανείς να εξετάσει αυτή την πτυχή ε, σχετικά με τις διάφορες ε, προδιαγραφές. Γνωρίζετε μη τη συζήτηση η οποία διεξάγεται εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι υπάρχουν δηλαδή ορισμένες προδιαγραφές οι οποίες δεν είναι διαπραγματεύσιμες δηλαδή όταν πρόκειται για την ασφάλεια των τροφίμων δεν θα μειώσουμε ε, τις απαιτήσει μας για την είσοδο στην ευρωπαϊκή αγορά. Δεν θέλουμε να μειώσουμε ε, αυτές ε, τις εγγυήσει, αλλά όταν πρόκειται για εργασιακά ή, περιβαλλοντολογικά θέματα υπάρχουν ορισμένα όρια στο τι μπορούμε να ζητήσουμε από τους εμπορικούς ομολόγους μας και χωρίς να αναφερθώ σε αυτή την αρνητική πτυχή θα ήθελα απλώς να σας πω ότι ουσιαστικά μια τέτοια συνεργασία σαν αυτή που έχουμε στο Μαρόκο είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς μπορούμε να εξετάσουμε αυτά τα διάφορα θέματα του περιβάλλοντος, της σημάνσεως στα πλαίσια συγκεκριμένων επιτροπών για να υπάρξει καλή συνεργασία και να τους υποκινήσουμε να εξυγχρονίσουν ορισμένες πτυχές και της αλληλείας τους. Παραδείγματο χάρη, σαν παράδειγμα θα μπορούσα να αναφέρω ότι το 2009 το Μαρόκο κατήρτισε ένα πρόγραμμα μέχρι το 2020 το οποίο μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο και συμμετέχουν στην ολοκληρωμένη ναυτιλιακή πολιτική της περιοχής συνεργαζόμαστε θαυμάσια στα θέματα της ασφαλείας των τροφίμων και τώρα έχουν πρόσβαση εις ορισμένα συστήματά μας υπάρχει ένας εκτενής φάκελος επ' αυτού υπάρχουν πολλά θέματα και εάν ουσιαστικά εστιαστώ εις την αλευτική πτυχή ε, του φακέλου και ήμουν ε, η Επιτροπή Αλληλείας ουσιαστικά θα ήμουν ικανοποιημένος με τα επιτεύγματα της ε, συνεργασίας με το Μαρόκο και αντιλαμβάνομαι ότι έχετε ανησυχίε για την εδαφική πτυχή και από αυτού θα δώσω το λόγο στον τον ομόλογό μου από την αρμόδια υπηρεσία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε εκπροσωπώ την Εξωτερική Επιτροπή Εξωτερικής Δράσεως και θα συμπληρώσω την απάντηση όσον αφορά την εδαφική πτυχή της εμπορικής συμφωνίας. Καταρχήν πρέπει να αναφερθώ στην επιστολή την οποία η κυρία Άστον και οι τρεις επίτροποι απίφθηναν εις τον πρόεδρο της Επιτροπής Ίντα το Μάιο όπου έδιδε από κοινού η Επιτροπή Εξωτερικής Δράσεως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μία απάντηση σχετικά με τα εδαφικά θέματα και τα οποία ανέπτυξα τον Ιούλιο στην Επιτροπή Ίντα. Η συμφωνία αυτή συνάδει με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στα θέματα του εμπορίου στις σχέσεις με το Μαρόκο. Πρόκειται για συμφωνίες που είναι ε, κατηρτισμένες από πολύ καιρό και θέλουν να προωθήσουν τις σχέσεις μεταξύ Μαρόκου και Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Οπότε η εμπορική συμφωνία σχετικά με τα γεωργικά και αληφτικά προϊόντα δεν αλλάζει ε, το σκηνικό και δεν προσθέτει νέα στοιχεία, απλούστατα διευκολύνει ε, εμπορικά ε, ορισμένες διαδικασίες και όσον αφορά το εδαφικό θέμα, όπως εξηγεί ξεκινήσαμε σε την επιστολή του Μαΐου θεωρούμε ότι η συμφωνία αυτή ε, συνάδει με τις διεθνείς συμφωνίες διότι το Μαρόκο σαν ε, μία δύναμη η οποία ε, εξασκεί η κυριαρχία ή στη Δυτική Σαχάρα δεν εκμεταλλεύεται τους πόρους της περιοχής και οι αρχές οι οποίες προβλέπονται όσον αφορά τα ωφέλη και τα συμφέροντα της της ε, τοπικής κοινωνίας δεν παραβιάζονται. Θεωρούμε λοιπόν ότι υπάρχουν διαβουλεύσεις και αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε ένα μέσο στην ε, ε, Συμφωνία Συνδέσεως, μία αρμόδια υποεπιτροπή η οποία παρακολουθεί και επαληθεύει ε, την εφαρμογή αυτής ε, της ε, εμπορικής συμφωνίας. Βεβαίως οι ομόλογοι μας συμφωνούν να μας δώσουν όλες τις πληροφορίες για την εφαρμογή της συμφωνίας και θα μπορέσουν οι υπηρεσίες να μεταβιβάσουν αυτές τις πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως γινόταν πάντα. Όσον αφορά λοιπόν την εδαφική πτυχή δεν υπάρχει νέο στοιχείο, δεν υπάρχει αλλαγή της νομικής καταστάσεως η οποία αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά απλώς πιο ευνοϊκά εμπορικά ε, ε, ε, τιμολόγια. Επίσης η ε, περιοχή αυτή δεν θα μπορούσε ε, να επωφεληθεί αυτών των δυνατοτήτων εάν εφαρμόζονταν αυτό που ζητάτε εσείς και ε, θα υπήρχε μια αρνητική επίπτωση. Αυτά είχα να πω όσον αφορά την εδαφική πτυχή. Ναι. Κύριε Ρωμέβα, έχετε το λόγο να πείτε ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ πολύ έχω μια αίσθηση ντεζοβή. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο επαναλαμβάνεται συνεχώς, το συζητάμε συνεχώς και τελικώς δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από το βασικό πρόβλημα κατά με, δηλαδή να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε κατά πόσον τηρείται ή όχι και νομίζω ότι αυτό είναι το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, η τήρηση του διεθνούς δικαίου. Υπάρχουν κάποιες πτυχές στις οποίες ανέφερε και η συναδέλφη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πω εντάχει κάποια στοιχεία γιατί πιεζόμαστε και από πλευρά χρόνου. Η κυρία Μπαρέα έθιξε το κατά πόσον μας αφορά ή όχι το εδαφικό ζήτημα. Για μένα είναι προφανές ότι μας ενδιαφέρει. Δεν μπορούμε να υπογράψουμε μια συμφωνία ή να υποστηρίξουμε μια συμφωνία της οποίας ε, δεν τηρείται η νομική βάση. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να καθορίσουμε σαφώς κατά πόσον υπάρχει τήρηση ή όχι. και νομίζω ότι μα τα ανέφερε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επαναλήφθηκε και στι επιστολέ που αναφέρονται στην Επιτροπή Ίντα το ζήτημα είναι κατά πόσον έχει το κυρίαρχο δικαίωμα το Μαρόκο να ρυθμίσει τους πόρους και τη διαχείριση μιας περιοχής η οποία νομικώς δεν είναι αρμοδιότητά της. Υπάρχουν τρόποι για την επίλυση του ζητήματος αυτού. Ε, κάποιοι από τους τρόπους αυτούς ε, από πλευράς ε, διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής ε, δεν είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής μας, αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα μπορούσαμε να θίξουμε σε μια συμφωνία της μορφής αυτής. Θα αναφερθώ σε δύο θέματα ε, η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Νορβηγίας με το Μαρόκο για τις ελεύθερες εμπορικές συναλλαγές. Και η Νορβηγία και οι Ηνωμένε Πολιτείες δηλώνουν ρητός ότι στις ε, συμφωνίες τους αποκλείεται η περιοχή της Δυτικής Σαχάρας γιατί θεωρούν ότι το βασίλειο του Μαρόκου δεν είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των πόρων της Δυτικής Σαχάρας. Αυτό έχουμε προτείνει επανειλημμένως να γίνει και στις δικές μας συμφωνίες και αυτό εξακολουθώ να καταλαβαίνω γιατί δεν μπορεί μπορεί να το θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει προηγούμενο σε άλλες παρόμοιες συμφωνίες, συμφωνίες ελευθέρων εμπορικών συναλλαγών και Αποδεικνύεται λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και είναι για κάτι απαραίτητο κατά εμέ. Είναι ένας τρόπος για να επιλύσουμε τη συγκεκριμένη συζήτηση και να προσπαθούμε ε, ε, συνεχώς να λύσουμε το ίδιο ζήτημα. Όσον αφορά τώρα τις εγγυήσεις που μας προσφέρει το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Μαρόκου διαβουλεύεται με τις ενδιαφερόμενες πλευρές. Συγγνώμη, αλλά είναι ελάχιστες αυτές οι διαβουλεύσεις και ελάχιστε οι εγγυήσει, διότι ο μόνο ενδιαλεγόμενο που έχουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η κυβέρνηση του Μαρόκου. Και νομίζω ότι χάνουμε τη διάσταση του προβλήματος. Γι' αυτό και ακριβώς επιμένω ότι χρειάζεται μία γνώση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής των απόψεων και των θέσεων της άλλης πλευράς, ε, του, των Πολυσάριων σε αυτή την περίπτωση. Και εξακολουθώ να θεωρώ ότι δεν είναι ένα θέμα στο οποίο δεν έχει άποψη το μέτωπο Πολυσάριο. Ως προς την ουσία τώρα, αναφέρθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάποια στοιχεία όσον αφορά την ε, ουσία για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Το είπα και συμφωνώ ότι νομικός εδώ δεν προσπαθούμε να διευκρινίσουμε την προέλευση, αλλά με βάση τη συμφωνία μπορούμε να έχουμε την θεσία χωρίς να ε, παρανομούμε. Τηρούμε τους κανόνες. θα ήταν απαραίτητο, το θέτω έτσι δυνητικά, ε, να γνωρίζουμε την προέλευση των προϊόντων ε, και για υγειονομικούς ε, και για κοινωνικούς αλλά και για εδαφικούς λόγους γιατί καλό θα ήταν οι καταναλωτές να γνωρίζουν από ποιον προέρχονται αυτά τα προϊόντα. Δημιουργούνται αρκετά ερωτηματικά με την τρέχουσα συμπεριφορά και καλό θα ήταν να αλλάξει η στάση μας για να μπορέσουμε να έχουμε λύσεις και καλό θα ήταν να το θέσουμε εδώ το ζήτημα. Όταν έχουμε συμφωνία αυτών των χαρακτηριστικών, το γεγονό ότι μπορούμε να έχουμε απελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών, μπορούμε να έχουμε συνεργασία με την ε, τρίτη χώρα, αλλά υπάρχει περίπτωση να προκύψει και το αντίθετο. Αρκετοί παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μεταφέρουν τις επιχειρήσεις τους και έτσι, εάν υπάρχουν κάποιες ευελιξίες σε αυτές τη χώρα, να εξάγουν από εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντα τα οποία πληρούν λιγότερες απαιτήσει από αυτές που ζητούνται ε, όταν οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι γεγονός. Δεν το επινόησα εγώ αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να το έχουμε κατά νου όταν κάνουμε αξιολόγηση και βλέπουμε τα υπέρ και τα κατά αυτών των συζητήσεων. Δεν θα την κάνουμε βέβαια αυτή τη συζήτηση σήμερα. Γνωρίζουμε όλοι ότι πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να παρακολουθούμε στενά στις συζητήσεις στην αρμόδια επιτροπή και στις 22 Σεπτεμβρίου θα μπορέσουμε να ξαναδούμε και κάποια θέματα και να δούμε κατά πόσον έχουμε προχωρήσει και στα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ρωμέβα. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροφή στις 10... Συγγνώμη, θα το συζητήσουμε στις 19 ε, Σεπτεμβρίου και θα ψηφίσουμε και 22 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσει η αρμόδια Επιτροπή. Ολοκληρώνεται λοιπόν το θέμα 6 και περνάμε στο επόμενο σημείο. Αλληλευτικέ δυνατότητε και χρηματική αντιπεροχή που προβλέπονται στη Συμφωνία Αλληλευτική Σύμπραξη μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και του Βασιλείου του Μαρόκου. Παράταση κατά ένα χρόνο λοιπόν. Ο κύριος Χάγκλουντ είναι εισηγητής. Επειδή λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε τι θα συζητήσουμε, να δώσουμε απευθεία το λόγο στον κύριο Χάγκλον για να μας πει τις απόψεις του επί του ζητήματος. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτοί από εσά που είχαν την ευκαιρία να παρίστανται στη συνεδρίαση την οποία έγινε και κλεισμένων των θυρών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις αληφτικές συμφωνίες πριν το καλοκαίρι γνωρίζουν γιατί το θέμα αυτό επανέρχεται σήμερα προς συζήτηση και έχει ήδη συζητηθεί μία φορά και ακούσατε και τα σχόλια του συναδέλφου μου επί του θέματος αλλά για όσους από εσά δεν ήταν είναι παρόντες τότε. Θα επαναλάβω ορισμένα από τα θέματα αυτά και θα σας παρουσιάσω μία σύντομη επισκόπηση για το πώς αντιλαμβανόμαστε αυτή την έκθεση. Αυτοί από εσά οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει το θέμα αυτό θα ήθελα να σας πω ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες είχαν ενδιαφερθεί πολύ ε, για την ε, συμφωνία αυτή και πρέπει να σας πω ότι από την αρχή της θητείας είχαμε ε, ρωτήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να διαπραγματευτεί το, τη συμφωνία και το πρωτόκολλο με το Μαρόκο το είχαμε ρωτήσει πρώτη φορά το 2009 αν θυμάμαι καλά και πέρυσι το χειμώνα όταν η συμφωνία καθορίστηκε επειδή υπήρξε κάποια εξέλιξη η Επιτροπή ε, μας είπε από τόμος ότι είχαν αποφασίσει να παρατείνουν για ένα χρόνο το πρωτόκολλο. Ε, ήταν ε, μια διαδικασία στην οποία νομίζω ότι δεν είχε αντιμετωπιστεί σωστά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ορισμένοι από εσά το είχαν ε, ήδη θίξει τον Ιούλιο. Είχα καθοριστεί σαν εισηγητής και η έκθεση αξιολογήσεως η οποία είναι πολύ σημαντική για μας είχε προχωρήσει διότι είχαν περάσει τέσσερα χρόνια από τις αξι... τελευταίες και ε, το Δεκέμβριο δηλαδή ε, μετά την παράταση της συμφωνίας ε, Ε, διότι η συμφωνία ξέπνε τον Φεβρουάριο φέτος ε, υπήρχε μία έκθεση μόνο γαλλικά εγώ ανέλαβα την έκθεση αυτή δυστυχώς δεν μιλώ γαλλικά και ε, παρόλη την βοήθεια συναδέλφων όπως ο, ο, Καντέκ δεν ε, ε, προχώρησε αρκετά γρήγορα. Μιλώ τέσσερις ευρωπαϊκές γλώσσες ε, αλλά κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε ότι τα έγγραφα αυτά είναι εμπιστευτικά και δεν μπορούσε να μου τα δώσει. Επίσης είχε εντωμεταξύ αναθέσει την ε, έκθεση ε, αξιολογήσεως σε μια ε, εταιρεία συμβούλων και ε, δεν είχα έγγραφα γερμανικά πράγμα που θα, είχε, θα με είχε βοηθήσει τα πράγματα ήταν περίπλοκα ζήτησα μετά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν μπορούσα να έχω μία έκθεση είτε σουηδικά που είναι η μητρική μου είτε αγγλικά είτε γερμανικά μου είπαν όχι μετά ήρθα σε επαφή με την Επίτροπο την οποία γνωρίζω και σέβομαι πολύ η οποία κατάλαβε τη θέση μου, μου είπε θα λύσει το πρόβλημα και το έπραξε αλλά μου είπε ότι θα είχα γρήγορα την μετάφραση και χρειάστηκαν τρεις μήνες μέχρι ότου την παραλάβω. Ε, μετά λοιπόν από όλα αυτά τα διαβήματα και ε, τις πιέσεις προς ε, την Επίτροπο η οποία μου είχε υποσχεθεί τη μετάφραση και όλα αυτά ε, επηρέασαν τη κατάσταση διότι το Κοινοβούλιο όπως ξέρετε διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτές τις συμφωνίες και λυπούμε πάρα πολύ ότι η Επιτροπή ανέλαβε να παρατείνει τη συμφωνία χωρίς να μας συμβουλευτεί πράγμα το οποίο έπρεπε να έχει κάνει. Η έκθεση όμως αξιολογήσεως είναι πολύ σημαντική. Ξέρω ότι ε, λίγοι την έχουν διαβάσει, εγώ και κάποιοι συνάδελφοι, ε, ορισμένοι ε, ίσως το έπραξαν χθες ή προχθές, αλλά μέχρι τότε μόνο τρεις από εμά την είχαν δει και θέλω να θίξω ορισμένα θέματα τα οποία νομίζω ότι σας αφορούν. Αναφέρομαι εδώ ε, στα συμπεράσματα της εκθέσεως αξιολογήσεως όπου λέγεται ότι τα αποτελέσματα της ε, ε, πρώτης τετραετίας εφαρμογής της συμφωνίας με το Μαρόκο είναι μάλλον απογοητευτικά πράγμα το οποίο είναι περίεργο εφόσον παρατείνεται ένα πρωτόκολλο και δεν έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη της ε, αλληλευτικής αγοράς και στην σταθεροποίηση. Ε, επίσης ε, όσον αφορά τα διάφορα προγράμματα δια πιστώνουμε ότι οι, τα αλλιεύματα στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας είναι ε, απλώς ε, επουσιώδη ε, και συνεχίζει εντάχει ο μιλητής διαβάζοντας κάποιο κείμενο που δεν έχουν οι ότι η συμφωνία αυτή δεν είναι σημαντική διότι δεν συμβάλλει στην οικονομία του Μαρόκο και, και και ε, δεν έχει προσφέρει ιδιαίτερα ε, ε, προσόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χαμηλό το κόστος της εφαρμογής διότι δεν έχουν διαπραγματευτεί σημαντικά αλλιευτικά, σημαντικές αλλιευτικές δυνατότητες και το κόστος είναι ε, πολύ υψηλό σε σχέση με τα ωφέλη τα οποία αποκομίζει η Ευρώπη από αυτό και βρίσκεται ε, κάτω από τα επίπεδα άλλων πανεφερών συμφωνιών που έχει ε, πραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι τελειώνει η έκθεση αξιολογήσεως. Από όλες τις εκθέσεις ε, πιστεύω ότι η έκθεση αυτή είναι πολύ ε, βαριά ε, για τους Ευρωπαίους φορολογουμένους είναι η λιγότερο επιτυχής από όλες τις ε, αλλιευτικές διμερείς συμφωνίες ε, που έχει διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα όλα αυτά δεν είναι πολύ θετικά. Ε, θα προσπαθήσω να καταρτήσω μία ικανοποιητική έκθεση κοιτάζοντας και τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν από πολιτική σκοπιά και Αυτά είναι τα στοιχεία που είχα. Από πλευρά οικολογική που επίσης μα ενδιαφέρει, αν κοιτάξουμε τα αποθέματα των 11 των 11 ε, ειδών που ψαρεύονται εις ε, το, εις Μαρόκο ε, στα πλαίσια των βυθικών ειδών η δεν έχουμε συμβάλει στην ανάπτυξη του τομέα αυτού της αλληλείας του Μαρόκο και ε, θα πρέπει να στηρίζουμε υπεύθυνες ε, αλευτικές πρακτικές πράγμα το οποίο τα τεχνικά δεν γίνεται στο Μαρόκο και εδώ απλώς διαβάζω τα πορίσματα ε, των συμβούλων. Όλα αυτά λοιπόν με ανησύχησαν και ιδίως με με ανησύχησε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα γνώριζε όλα αυτά τον Δεκέμβριο και παρόλα αυτά αποφάσισε να παρατείνει το πρωτόκολλο για ένα χρόνο πράγμα το οποίο δεν είναι σωστή διακυβέρνηση και ε, χρηστή χρήση των ε, πόρων των φορολογουμένων. Ε, ζήτησα λοιπόν από την Επιτροπή και τον Επίτροπο, την Επίτροπο να μου πούν τι σκοπεύουν να κάνουν και ε, έκτοτε έχει περάσει άλλος ένας χρόνος διότι ε, δεν θα ολοκληρώσουμε την εξέταση του θέματος ε, μέχρι τον Οκτώβριο και θα είμαστε πολύ κοντά στην ημερομηνία του, Φεβρουαρίου, του επόμενου Φεβρουαρίου και εντωμεταξύ μεταξύ προέκυψε και το θέμα της Δυτικής ε, Σαχάρας όταν εξετάσουμε την γνωμοδότηση του συνάλφου Ρωμέβα. Πρέπει λοιπόν να δούμε αν είναι βιώσιμη αυτή η συμφωνία ε, νομικά ε, για αν εξετάσουμε την κατάσταση της Δυτικής χάρας. Σε όλα αυτά τα θέματα άλλωστε η έκθεση αξιολογήσεως δεν μας βοηθά και η ε, νομική επιτροπή έχει εκφραστεί διαφορετικά από από την, ε, τα σχόλια των εκπροσώπων της ε, Επιτροπής Εξωτερικής Δράσης που ακούσαμε προηγουμένως της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης που ακούσαμε προηγουμένως. Αυτές είναι οι πληροφορίες τις οποίες έχω στη διάθεσή σας. Πρέπει να πω ότι ε, τα θετικά σημεία ήταν ελάχιστα και θα ήθελα να είχαμε την ε, ευκαιρία να επισκεφθούμε το Μαρόκο, πράγμα το οποίο επιθυμούσαμε, αλλά ε, υπήρχαν, ε, υπήρξαν ορισμένα προβλήματα στις επικοινωνίες με τη μαροκινή πλευρά και η γραμματεία μας ποτέ δεν κατάφερε να τα ξεπεράσει γι' αυτό και όταν εγώ ρώτησα τον ε, την Άνοιξη ε, τι γίνεται μου είπαν ότι δεν ήξεραν ότι το Κοινοβούλιο ήθελε να επισκεφθεί το Μαρόκο. Αυτά είχα να σας πω και παρακαλώ όλους όσους ενδιαφέρονται για το θέμα να διαβάσουν την έκθεση αξιολογήσεως διατίθεται τώρα αγγλικά είναι ενδιαφέρουσα και τον Οκτώβριο θα χρειαστεί να λάβουμε μία απόφαση επί του θέματος και να προχωρήσουμε ε, στην επόμενη φάση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σκάτεκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητέ Κάλλη, εγώ δεν μιλάω φιλανδικά, ζητώ συγγνώμη, αλλά τι να κάνω. Παρόλα αυτά, ε, διαβάσαμε την ίδια συμφωνία, την ίδια έκθεση, αναρωτιέμαι, δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Νομίζω ότι το πρωτόκολλο 25 Ιουνίου 2011 που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συνάδει πλήρω με την εντολή που ανέθεσε το Συμβούλιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, τα πλήστα κράτη-μέλη υποστηρίζουν το πρωτόκολλο. Η Συμφωνία Εταιρική Σχέση έχει ιδιαίτερη σημασία κατά τη γνώμη μου. Σημαντικό για τον αλλιευτικό στόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε εμπορικό επίπεδο. Υπενθυμίζω ότι επιτρέπει σε 10 κράτη-μέλη να αλλιεύουν στα ε, ύδατα του Μαρόκου και βελτιώνει την την ποιότητα των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου γιατί είναι ένας βασικός εταίρος λόγω εγκύτητας ε, των ε, εδαφών μας. Όπως είπαμε και σε προηγούμενη έκθεση, Υπάρχει το πολιτικό πρόβλημα της Δυτικής Σαχάρας ε, που δημιουργεί διαστάσεις απόψεων και έντονες συζητήσεις στην Επιτροπή. Φυσιολογικό είναι αυτό. Ε, το έχω ξαναπεί αλλά το επαναλαμβάνω. Ε, δεν θα ρυθμίσει το πρόβλημα η Επιτροπή Αλίας. Δεν θα ρυθμίσει η Επιτροπή Αλίας ένα ζήτημα διεθνούς δικαίου. Ε, η Κατρίν Τροτμάν το είπε προηγουμένως. Ε, αυτό ε, είναι, αποτελεί αρμοδιότητα γενικότερα της διεθνούς κοινότητας και ο ΙΕ έχει επιληφθεί του ζητήματος. Ε, συμφωνώ ότι η διεθνής κοινότητα δεν επιδεικνύει ιδιαίτερο, ιδιαίτερη τόλμη, αν θέλετε, στην περίπτωση της Δυτική Σαχάρας. Εντάξει, δεν είμαστε ε, προτεργάτες, ε, συμφωνώ, αλλά ο μοναδικός ε, συνομιλητή μας σήμερα, νομικός πώ είναι το βασίλειο του Μαρόκου και δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Δεύτερον, συγγνώμη γιατί μπερδεύτηκα. Η κυβέρνηση του Μαρόκου υιοθέτησε εθνική στρατηγική στον τομέα της αλίας, χάρη στην οποία δημιουργήθηκαν 42.000 νέες θέσεις απασχόλησης, δεν είναι αμεληταίο, 21.000 ε, από αυτές. Βάσει των στοιχείων που έχω στη διάθεσή μου, έτσι, δημιουργήθηκαν στον Νότο, στη Δυτική Σαχάρα, εν προκειμένου. Νταρλά, Λαγιούν και τα λοιπά, σε όλα αυτά τα λιμάνια. 200.000 ευρώ έχουν επενδυθεί σε προγράμματα ανάπτυξης του αληφτικού κλάδου στην περίοδο 2007-2011, δεν είναι αμελητέο, Στη Δυτική Σαχάρα 44 εκατομμύρια ευρώ διοχετεύθηκαν σε προγράμματα που αποσκοπούν στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Προτείνω λοιπόν να πάμε επί τόπου, να διαπιστώσουμε όλα αυτά τα έργα που έχει αναλάβει και έχει φέρει σε πέρας η κυβέρνηση του Μαρόκου, ας πάμε επιτόπου να δούμε τι έχει γίνει με αυτές τις επενδύσεις, γιατί αυτές οι επενδύσεις είναι υποφελεί για την Μαροκινή Αλία και για τους Σαχράουι. Δεν ε, ε, ε, και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και Μαροκινοί, όχι μόνο Σαχράοι που διαβίουν στη Δυτική Σαχάρα. Υπάρχει και ένα νέο άρθρο που προβλέπεται υποβολή ετησία έκθεση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη στήριξη του κλάδου, αυτό που σχολίασα δηλαδή, και σχετικά με τη γεωγραφική κατανομή αυτή τη υποστήριξη. Αυτό αποτελεί ηχέγιο κατά τη γνώμη μου. Άρα δεν βλέπω να υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτή τη συμφωνία. Νομίζω αντίθετα ότι είναι πάρα πολύ καλή αυτή η συγκεκριμένη συμφωνία. Ακριβή, ναι, ναι, ναι, κοστίζει χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ομολογώ αλλά ε, είναι σημαντική γιατί δεν δημιουργεί ουσιαστικά προβλήματα στα εμπλεκόμενα μέρη. Νομίζω ότι θα έπρεπε να ε, το αφήσουμε αυτό στην κρίση των αρμοδίων αρχών. Και πάλι θα πω ότι δεν διαβάσαμε ε, τι ίδιε εκθέσει ή δεν ερμηνεύσαμε ε, με τον ίδιο τρόπο τα αριθμητικά στοιχεία, γιατί είμαι από αυτού, ε, στου οποίου αναφερθήκατε, που διάβασαν όντω αυτή την έκθεση για το Μαρόκο, αλλά δεν την ερμηνεύσαμε με τον ίδιο τρόπο. Εγώ αυτά πιστεύω. Σα ευχαριστούμε, κύριο Δρομέρα. Ε. Ναι. Προφανώς υπάρχει σχέση με την προηγούμενη συζήτηση, αλλά υπάρχουν φυσικά και ίδια στοιχεία της συγκεκριμένη ε, συζήτησης. Επιμένω λοιπόν ότι είναι λίγο διαφορετικό το πλαίσιο από την προηγούμενη συζήτηση. Εδώ έχουμε ένα πρωτόκολλο συμφωνίας, το οποίο αφορά συγκεκριμένα τους αλλιευτικούς πόρους μιας περιοχής. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι μόνο το Μαρόκο, αλλά επικουρικά περιλαμβάνουν και κάποια ε, χωρικά είδητα τα οποία είναι υπό ή υποσυζήτηση, για να είμαι λίγο πιο ήπιες. Τα θέματα τα οποία έθιξε ο κύριος Κλάντ είναι σημαντικά και θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Καταρχάς, το είπε σαφέστατα άλλωστε ο κύριος Χάγκλουντ, αλλά και ανησυχητικά, είναι το θέμα των αποθεμάτων. Η πρώτη ανησυχία λοιπόν που έχουμε είναι τα αποθέματα. Διάβασα και εγώ την ε, συγκεκριμένη έκθεση και αντιλαμβάνουμε ότι πρόκειται για ένα στοιχείο το οποίο θα έπρεπε από μόνο του να μας ανησυχήσει ιδιαίτερα. Δεύτερον, ο οικονομικός παράγων δεν είναι κάτι ίσονος σημασία και εδώ νομίζω ότι διαφωνώ εν μέρη με τον συνάδελφο Καντέκ διότι αν είναι σωστά τα αριθμητικά στοιχεία και δεν έχω κανένα λόγο να τα αμφισβητήσω, είναι απαραίτητο όχι μόνο να γνωρίζουμε, αλλά και να εξηγήσουμε ότι αυτή η συμφωνία δημιούργησε κάποιες απώλειες ε, πολύ σημαντικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η πιο συγγνώμη, είναι η λιγότερο προσοδοφόρα οικονομικά συμφωνία από αυτές που είχαμε με διάφορα μέρη του κόσμου. Είχαμε μόνο 0,86 σεντ για κάθε ευρώ το οποίο καταβάλαμε από τα 36 εκατομμύρια ευρώ που κατέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση για, το, ε, για τη συμφωνία αυτή. Πρόκειται λοιπόν για κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτούμε ιδιαίτερα. Το τρίτο στοιχείο είναι το νομικό στοιχείο. Δεν ε, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτό το φαύλο κύκλο και από αυτή τη συζήτηση όπου κάποιοι θεωρούν ότι είναι νόμιμο, κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι είναι απαράνομο, κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι ανταποκρίνεται στην ε, νομιμότητα, κάποιοι άλλοι θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνεται. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι προασπίζονται και εγώ επιμένω σε αυτό το γεγονός ότι η Δυτική Σαχάρα δεν αποτελεί τμήμα του Μαρόκου, επομένως το βασίλειο του Μαρόκου δεν μπορεί να διαχειρίζεται τα αποθέματα της Δυτικής Σαχάρας, αλλά ούτως ή άλλως κάποιοι συνάδελφοι εξημών θεωρήσαμε ότι ήγηκε η ώρα να φτάσουμε ε, με το θέμα αυτό στο ε, δικαστήριο. Και νομίζω ότι θα πρέπει να κινητοποιηθούμε περισσότερο τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες εβδομάδες, διότι όπως προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας και όπως έχουμε κάνει και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, άπτεται πλέον στο δικαστήριο να καθορίσει κατά πόσον αυτό το πρωτόκολλο τηρεί τα όσα περιλαμβάνουν οι συνθήκες και το διεθνές δίκαιο και αν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε, που είναι να ασχολούμαστε με ένα θέμα ε, που αφορά την Επιτροπή Αλληλείας ε, και δεν έχει επιληθεί σε διεθνές επίπεδο. Εξακολουθούμε να λέμε ότι εμείς ως Επιτροπή Αλληλείας δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να καθορίσουμε την κατάσταση. Αυτό που θέλουμε όμως εμείς είναι να πάει απευθείας το θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να καθορίσει κατά πόσον είναι νόμιμο ή όχι αυτό το πρωτόκολλο και φυσικά αυτό θα μας διευκολύνει ιδιαίτερα για τις επόμενες συζητήσεις οι οποίες έχουν σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Οι συνθήκες είναι αυτές που γνωρίζουμε όλοι και νομίζω ότι για την έκθεση του κυρίου Χάγκλαντ θα υπάρχουν άμεσες επιπτώσεις. Μπορούν να είναι δύο παραλλήλου διαδικασίες άλλωστε. Δεν υπάρχει και μεγάλη ανάγκη να ε, είναι αλληλένδετης απαραίτητα. Πρέπει όμως να περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου για να δούμε κατά πόσον το ε, Κοινοβούλιο θα λάβει απόφαση για την ανανέωση αυτής της συμφωνίας. Ο κύριος Στίβενσον. Ευχαριστώ να συγχαρώ τον Καρλ Χάγκλουν πρώτα απ' όλα γιατί εργάστηκε πάρα πολύ σκληρά. Ενημέρωσε ολόκληρη την Επιτροπή για ε, σειρά ζητημάτων που αγνοούσαμε, έτσι, τουλάχιστον πολλοί από εμά. Ε, και πρωτήτερα ήμουν μάλλον υπέρ ε, τη συνέχιση αυτή τη συμφωνία Δηλαδή αν αποσυρθούμε ε, θεωρούσα ότι το Μαρόκο θα πολλούσε τα δικαιώματα αλλία σε χώρες που δεν ασχολούνται με πόσοι Σαχράου βρίσκουν δουλειά στη Δυτική Σαχάρα, δεν ασχολούνται με περιβαλλοντικά πρότυπα, δεν ασχολούνται με την ε, εξάντληση των αλλιευτικών αποθεμάτων και έτσι θα επιδεινωνόταν περαιτέρω η κατάσταση και εγώ θεωρούσα ότι άξιζε τον κόπο παρότι είναι δαπανηρή συμφωνία θεωρούσα ότι άξιζε να συμβάλλουμε κατά αυτόν τον τρόπο να δώσουμε κάποια από τα χρήματα των φορολογουμένων, ούτω ώστε να προστατεύσουμε την Δυτική Σαχάρα, να ε, αποτρέψουμε την υπεραλίευση. Αλλά από όσα ακούω τώρα από τον κύριο Χαγκλούντ, ε, βλέπω ότι εξαντλούνται τα αποθέματα βενθικών ειδών, δηλαδή σχεδόν όλα τα βενθικά είδη υπεραλλιεύονται, δεν γίνεται σωστή ανάλυση. Ε, οικονομικά ε, αυτό έχει ε, καταστροφικές επιπτώσεις και με σοκάρει ο τρόπος που, με τον οποίο χειρίζεται το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πραγματικά δεν κινείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών της συνθήκης της Λισαβόνας. και όταν ο εισηγητής αυτή μα προσπάθησε να μιλήσει με την ίδια την Επίτροπο για να υπερβούμε αυτά τα προβλήματα ε, και ε, προσπάθησε να συνεννοηθεί με τη γραμματεία και δεν τα κατάφερε. Νομίζω ότι αυτό είναι απαράδεκτο και ελπίζω όλοι να αντλήσαμε ένα χρήσιμο δίδαγμα από αυτήν την έλλειψη ε, εφαρμογή τη διαθεσμική συμφωνία και να ληφθεί αυτό υπόψη μελλοντικά όταν θα μα αποσχολήσουν και άλλε τέτοιε συμφωνίε. Έχοντα ακούσει τώρα την παρουσίαση τη έκθεση από τον κύριο Χάγκλουντ, ε, θυμάμαι ότι και σε προηγούμενε συνεδριάσει είχα μιλήσει για δύο μεγάλε σκοτσέζικε στράτε που είχαν εμπλακεί στην ε, αλληλεία αυτών των υδάτων και οι πλειοκτήτε που αλλιεύουν στη Δυτική Σαχάρα ε, είχαν απασχολήσει 6.000 Σαχράουι ε, σε ένα εργοστάσιο μεταπίεσης και εκφορτώνουν στη Δυτική Σαχάρα όλα τα αλλιεύματά τους. Αναφυσβήτητα λοιπόν ο λαός της Σαχάρα δεν πρόκειται εμείς, δεν πρόκειται να υποφεληθεί αν εμείς αποσυρθούμε από τη συμφωνία αυτή διότι η κυβέρνηση του Μαρόκου δεν ενδιαφέρεται για το ποιος θα απασχοληθεί αρκεί το κράτος να μπορέσει να έχει τα έσοδα από οποιονδήποτε, από τους Ιάπωνες ή οποιονδήποτε άλλο. Εάν λοιπόν αποβλέπουμε ή στο να στηρίξουμε αυτή την συμφωνία συνεργασίας θα πρέπει να βρουν ένα καλύτερο τρόπο να το αποδείξουν. Ο κύριος Σάντσες Πρισέδο. Ναι, συγγνώμη. Αφαιρέθηκα λίγο. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον εισηγητή και την παρουσίασή του και για τα όσα έκανε. Νομίζω ότι έθιξε μια σειρά από ανησυχίες, όπως είπε και ο κύριος Ρομέδα, οι οποίε είναι καθόλου ένομες. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ δύο κατηγοριών. Καταρχάς τα βραχυπρόθεσμα μέτρα και κατά δεύτερον τα μακροπρόθεσμα ζητήματα. Τα βραχυπρόθεσμα είναι η παράταση αυτής της αλληλευτικής συμφωνίας για το τρέχον έτος και σε περίπτωση που διακοπούν οι αλληλευτικές δραστηριότητες θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν πολύ αρνητικέ συνέπειες για το στόλο μας, για περιοχές οι οποίες ε, πλήττονται ήδη από την ε, οικονομική κρίση και ε, επομένω, και ο πληθυσμός πλήττεται από την οικονομική κρίση η Δυτική Σαχάρα στη συμφωνία δεν αναφέρεται σε κυριαρχία, αναφέρεται σε χωρικά ύδατα και σε ύδατα της δικαιοδοσίας ε, του Μαρόκου. Κάποιες από τις ανησυχίες επιτροπές ε, ήταν ε, οι επιπτώσεις για τη Δυτική Σαχάρα και νομίζω ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ σαφής διότι λέει ότι στις 13 Δεκεμβρίου νομίζω είχαμε ε, για πρώτη φορά πληροφορίες και οι πληροφορίες αυτές αποδεικνύουν ότι ε, την περιοχή διότι δημιουργούνται θέσεις εργασίας και υπάρχουν και κάποια επιπλέον έσοδα. Αυτά λοιπόν ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα. Υπάρχουν όμως ένα, κάποια πιο συνολικά θέματα που αφορούν το τι μέλη γενέστε, τι θα κάνουμε στο μέλλον και τι όρους πρέπει να έχουμε, οι οποίοι κατά την άποψή μου πρέπει να διατηρηθούν για να μην έχουμε επιπλέον προβλήματα αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, τι μπορούμε να έχουμε για να έχουμε μια ισορροπημένη αλληλευτική συμφωνία και νομίζω ότι σε αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Θεωρώ ότι η ανάλυση κόστους ωφελίας δεν είναι απλώς μια ανάλυση που αναφέρεται μόνο στις αλληλευτικές δυνατότητες. Αν θέλουμε να κάνουμε μια εμπορική συναλλαγή δεν θα πρέπει να σταθούμε μόνο στην αλληλευτική συμφωνία, να δούμε, θα μπορούμε να δούμε τις τιμές και να κάνουμε μια σύγκριση. Μια αλληλευτική συμφωνία είναι κάτι επιπλέον, δεν είναι μια απλή εμπορική συμφωνία, είναι μια συμφωνία που μας επιτρέπει... Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ω αλληλευτικός παράγων σε διεθνέ επίπεδο να συνεισφέρει στην ανάπτυξη τη αλληλεία και σε άλλε χώρε. Ε, και Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καθορίσει μια στρατηγική συμφωνία που θα μας επιτρέψει ε, να έχουμε καλύτερες αλληλευτικές δυνατότητες. Υπάρχει λοιπόν αξία και ως προς αυτό και αυτή η αξία αποτελεί τμήμα των ελευτικών συμφωνών, διότι οι ελευτικές συμφωνίες έχουν επιπτώσεις και στη συγκεκριμένη επικράτεια με την οποία συνάπτεται η συμφωνία και θα πρέπει να δούμε και πέραν λοιπόν των εμπορικών συναλλαγών. Υπάρχουν και αυτές οι πτυχές που ορισμένες φορές αγνοούμε. Και υπάρχει και κάτι ακόμα στο οποίο θα ήθελα να σταθώ, το θέμα της Σαχάρας. Νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να απαντήσουμε στα προβλήματα της Σαχάρας στις αλληλευτικές συμφωνίες. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την άγουσα. Αλλά αν θέλουμε να κάνουμε μια συνολική ανάλυση, θα πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε και οποιαδήποτε απόφαση επί του ζητήματος εάν προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ακόμα και το γεγονός ότι συμφωνούμε ότι η ε, διένεξη αυτή θα πρέπει να επιληθεί σε διεθνέ επίπεδο. Προσέξτε όμω, υπάρχουν διάφοροι τρόποι επίλυση ενό προβλήματο. και σίγουρα δεν θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τα προβλήματα και να δημιουργήσουμε και άλλα προβλήματα και να δημιουργήσουμε προβλήματα για την περιοχή που πλήττεται και να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν νέε δυνατότητε ανάπτυξη. Ο σωστό δρόμο λοιπόν είναι να προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα τα μικρά, τα οποία αφορούν του πολίτε καθημερινά και μετά να δούμε τι γίνεται με τα μεγαλύτερα. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το, ε, την θαυμάσια εργασία την οποία έχει κάνει και για την καλή σύνοψη ε, της εκθέσεως αξιολογήσεως. Εγώ διάβασα μόνο την περίληψη μέχρι στιγμής και αυτή ήταν διαθέσιμη αγγλικά και δεν ε, μπορεί κανείς να πει πολλά θετικά για τη συμφωνία αυτή από οποιαδήποτε οπτική γωνία είτε πρόκειται για σωστή ε, χρήση ε, χρημάτων ούτε για την, τα πλεονάσματα των αποθεμάτων διότι κάθε συμφωνία αλλιευτική πρέπει να βασίζεται σε αυτό το πολύ βασικό γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πλεόνασμα αποθεμάτων τα οποία αλλιεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ όλα τα αποθέματα ήδη υπεραλλιεύονται και υπάρχει μείωση σε ορισμένα είδη ψαριών. Δεν αναφέρω αναφέρομαι μόνο στα βυθικά είδη αλλά και στα πελαγικά είδη. Το μόνο πλεόνασμα ε, είναι ε, η Σαρδέλα στο νότο, δηλαδή στην περιοχή της Σαχάρας. Αλλά φαίνεται ότι όλα τα ίδια ήδη και ακόμη και στα σύνορα με την Μαυριτανία και άλλες χώρες δεν φαίνεται να υπάρχουν επαρκή αποθέματα. Πρέπει ενδεχομένως τα αποθέματα να ε, έχουν μετακινηθεί και υπάρχει και στην Κάμπια και στο Μαρόκο υπεραλίευση. Οπότε εγώ δεν νομίζω ότι μπορούμε να αυξήσουμε την αλίευση αυτών των ε, ειδών. Ε, μπορεί να υπάρχουν ε, θαλάσσια, θαλάσσια θηλαστικά τα οποία επίσης αλίευονται καθώς επίσης και καρχαρίες και όλα αυτά μας δημιουργούν ανησυχίες. Το Μαρόκο βέβαια έχει τη δυνατότητα να πουλά πόρους αλλιευτικούς που ανοίγουν ε, στα εδάφη της ε, Δυτικής Σαχάρας. Αυτό είναι ένα θέμα ε, το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ σοβαρά, ιδίως σε φέτος, με όλα τα γεγονότα τα οποία έχουν ξεσπάσει στην Βόρεια Αυτική. Βέβαια το Μαρόκο είναι ένας βασικός εταίρος μας και εμείς θεωρούσαμε ότι και η Τινησία και η Λιβύη και η Αίγυπτος ήταν σημαντικοί παράγοντες αλλά το θέμα είναι ποιος είναι πιο σημαντικός και η κατάσταση όντως γίνεται ε, πάρα πολύ δυσχερής ε, για ε, ορισμένες δικτατορίες και η πρόταση του κυρίου Ρωμέβα είναι η μόνη λογική διότι θα πρέπει να μπορέσουμε να λύσουμε το θέμα και να γνωρίζουμε αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η Δυτική Σαχάρα είναι μία περιοχή του Μαρόκου και αν το Μαρόκο μπορεί να πουλά τους φυσικούς πόρους αυτής της περιοχής γιατί ναι μεν οι αρχές του Μαρόκου προσφέρουν ε, χέγγια ότι όλα, τα, όλα αυτά είναι προς όφερον της ε, περιοχής της Σαχάρας αλλά μιλάμε για ένα καθεστώς στο Μαρόκο το οποίο ενδέχεται να μην επιβιώσει πέραν των έξι μηνών. Άρα η κατάσταση είναι πολύ περίπλοκη και συμφωνώ ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι το κατάλληλο, ε, ο κατάλληλος χώρος όπου θα πρέπει να κριθεί το θέμα αυτό. Ε, δεν ε, μπορούμε εμείς να κρίνουμε γιατί ακόμη και τα ψάρια είναι πολιτική. Πρόκειται για διατροφή, πρόκειται για τρόπο επιβίωσης δημοκρατική ε, διαδικασία και όλα, όλες αυτές οι πτυχές είναι σημαντικές. Γι' αυτό και θα συμφωνούσα ότι αυτό πρέπει να παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ε, με εκπλήσει ότι προηγουμένως ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απάντησε στην ερώτησή μου για τη διαφορά μεταξύ των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Ισραήλ σχετικά με τη διοικητική όχθη και των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την Σαχάρα με το Μαρόκο. Και γιατί δεν μου απαντήσατε πιο σαφώς. Η κυρία Ανδρές Παρέα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχουμε το ίδιο πρόβλημα που συζητήσαμε και προηγουμένω. Ευχαριστώ τον κύριο Χάγκλοντ για τι εξηγήσει που μα έδωσε, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε και πότε ακριβώς γίνεται αυτή η παράταση. Πρόκειται για μια παράταση, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι τα στοιχεία τα οποία της έδωσε το Μαρόκο επαρκούν ή δεν επαρκούν, δεν της δίνουν επαρκείς ε, εγγυήσεις και επομένως ζητά παράταση για να εξετάσει την κατάσταση. Μας είπατε κάποια πολύ αρνητικά στοιχεία και πρέπει να τα λάβουμε υπόψη αλλά θα μπορούσαν να μας χρησιμεύσουν για να καθορίσουμε τη νέα συμφωνία. Καλό είναι να εξετάσουμε τι συνέβη στο παρελθόν για να δούμε γιατί υπάρχει παράταση και να δούμε και ποια θα είναι τα κριτήρια για το μέλλον. Θεωρώ ότι θα πρέπει να καθορίσουμε περιβαλλοντικά μέτρα, εάν υπάρχουν όντως αυτές οι ελλείψεις, γιατί αξιολογήθηκαν, πώς αξιολογήθηκαν, με ποια κριτήρια. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία θα πρέπει να γνωρίζουμε για να δούμε ε, τι θα ευνοήσει και την αλληλεία. Όσον αφορά τώρα τη Συμφωνία Σύνδεσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, κάποιες επιπλέον ευθύνες, οι οποίες δεν είναι απευθείας αλλιευτικές είναι η βοήθεια και η ανάπτυξη του στόλου. Το Μαρόκο κάνει τη διαχείριση των ε, χωρικών υδάτων της ε, Σαχάρας, τα οποία γίνεται αλίευση αυτή τη στιγμή και θα πρέπει μέσω της συμφωνίας να υπάρξει και ανάπτυξη για τη συγκεκριμένη περιοχή και δημιουργία θέσεων εργασίας. Νομίζω ότι το να παρατείνουμε μια ε, κατάσταση τορπιλίζοντάς της κιόλα ε, κατά κάποιο τρόπο θα δημιουργήσει πολύ αρνητικές συνέπειες για την περιοχή. Η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μου φαίνεται ότι είναι κάτι σωστό. Νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσει να εργάζεται, να συνεχίσει να ε, βοηθά στη δημιουργία καλών συμφωνιών, οι οποίες θα είναι όχι μόνο προς όφελος του ελευτικού τομέα, αλλά και του ίδιου του πληθυσμού μιας περιοχής. Πρόκειται λοιπόν για ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που μας δίδεται αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια παράταση που μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε και να δούμε τι ε, ε, συμπεράσματα ή εξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από αυτή τη συμφωνία. Ε, η πρόεδρο, Θα πω και εγώ κάποια πράγματα τώρα. Έχουμε την παράταση αφενός ε, που προσπαθούμε να δούμε κατά πόσον θα την εγκρίνουμε ή θα την απορρίψουμε. Ε, εμένα θέμα, το θέμα της παράτασης, να σας πω την αλήθεια, λίγο με ανησυχεί. Αυτό που είναι αλήθεια και σε αυτό που έχει δίκιο ο κύριος Χάκλοντ είναι ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ επικριτική για την αλληλευτική συμφωνία με το Μαρόκο. Νομίζω ότι είναι η πιο αρνητική συμφωνία που έχω δει σε όλη τη ζωή μου από όλε τι εκθέσει αξιολόγηση που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ τη διάβασα από την αρχή μέχρι τέλου. Νομίζω ότι είναι η πιο επικριτική έκθεση που έχω διαβάσει εγώ. Υπάρχουν ε, ίσω και κάποια σημεία που μπορεί να είναι απόλυτα σωστά, αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ αρνητικά από τα όσα διάβασα σε αυτή την έκθεση. Καταρχάς, με τα όσα γνωρίζουμε για το θέμα της ελευτικής συμφωνίας ε, ε, με το Μαρόκο, Νομίζω ότι αυτό το οποίο ενδιαφέρει εμένα ουσιαστικά αυτή τη στιγμή και είναι κάτι το οποίο δεν ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ποια είναι η μελλοντική στρατηγική μετά από τις 28 Φεβρουαρίου που θα εκπνεύσει αυτή η συμφωνία. Και εδώ υπάρχουν δύο εναλλακτικέ λύσει. Ή συμφωνία ή μη συμφωνία. Εάν υπάρξει συμφωνία θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τον αλληλευτικό τομέα εκεί. Ε, εάν δεν γίνει συμφωνία θα πρέπει να γίνει σίγουρα επί άλλων βάσεων, τελείω διαφορετικών από αυτέ που έχουμε αυτή τη στιγμή. εκμεταλλεύεται τη συμφωνία ο μεγαλύτερο αριθμό του στόλου με την εξαίρεση του πελαγικού στόλου και πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ ακριβή ε, συμφωνία. Πληρώνουμε 30 τόσα εκατομμύρια ευρώ ε, από το σύνολο των 160 εκατομμυρίων ευρώ που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω είναι σχεδόν το 1 τρίτο των όσων πληρώνουμε για τι συμφωνίε. Θα πρέπει λοιπόν να τα κάνουμε όλα επί άλλη βάσεω. Αυτό που με ανησυχεί κύριε Χάντλουγκλουντ, διότι εσεί μιλάτε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ποια είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από την παράτηση της συμφωνίας. Ούτε η κυρία Δαμανάκη ούτε κανένας άλλος δεν μας ενημέρωσε. Και αυτό με ανησυχεί εμένα ιδιαίτερα διότι πρέπει να δώσουμε και μια απάντηση στον αλληλευτικό τομέα είτε υπάρχει συμφωνία, είτε δεν υπάρχει συμφωνία, είτε είναι τελείω διαφορετική συμφωνία, ο αληφτικό τομέα έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποιο θα είναι το μέλλον του. Διότι είναι αυτό ο τομέα που θα πρέπει να συνεχίσει να πληρώνει του υπαλλήλου του, που θα πρέπει να πληρώνει κοινωνικέ ασφαλίσει και θα πρέπει να έχουν ένα ελάχιστη δυνατότητα προγραμματισμού. Και δεν μπορούμε να είμαστε έρμεο των όσων θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Κοινοβούλιο. Πρέπει να του ενημερώνουμε εγκαίρω. Είτε θα υπάρξει είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία και αν υπάρξει τι θα γίνει με είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι δεν υπάρχει σαφήνεια από καμία πλευρά. Θα μιλήσω τώρα και για τη θεσμική πτυχή, στην οποία αναφέρθηκε και ο κύριος Χάγκλουντ. Υπάρχει το θέμα της ενημέρωσης. Εξακολουθούμε να μην μπορούμε να επιλύσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα της εμπιστευτικότητας των εκθέσεων αξιολόγησης. Εξακολουθούν να μας θέτουν παγίδες συνεχώς και ε, εμείς κάναμε πάρα πολλές προσπάθειες, εγώ ακόμα και με την κυρία Δαμανάκη έκανα συζητήσεις επί του ζητήματος και λύση καμία. Υπάρχει για παράδειγμα το θέμα της αξιολόγησης Γρυλανδίας τι έλεγε εμπιστευτικό. Χωρί καμία άλλη διασφάλιση, η Γρυλανδία είναι εμπιστευτική. Δεν ξέρω αν είναι στα αγγλικά ή στα γαλλικά, γιατί δεν την είδα. Εξακολουθεί να είναι εμπιστευτική αυτή η έκθεση. Με ενημέρωση γραμματέα ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο κύριο Μπούζεκ έλαβε μία επιστολή από τον κύριο Σέσκοβιτ, ο οποίο είναι αρμόδιο για όλα αυτά τα θέματα, ο οποίο τον παραπέμπει στην αναθεώρηση της Συμφωνίας Πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από εδώ και πέρα δεν θα δίνεται έγκριση σε κανέναν Ευρωβουλευτή για να παραστεί στις διμερείς συνεδριάσεις, στις συνεδριάσεις για τις διμερείς συμφωνίες. Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη, θα το συζητήσουμε άλλωστε και σε συνεδρίες των συντονιστών, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εκβιασμό άμεσο εκβιασμό και χρησιμοποιώ τον όρο εκβιασμό στα, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από εδώ και πέρα, διότι είναι απαράδεκτο κάθε φορά να καθυστερούμε λόγω των ίδιων προβλημάτων. Στην επόμενη συνεδρία των συντονιστών θα συζητηθεί το ζήτημα, αλλά θα ήθελα να γνωρίζετε ο κύριος Σεύκοβιτς απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος λέει ότι από εδώ και πέρα δεν δέχονται κανέναν ευρωβουλευτή ω παρατηρητή στις διμερείς συμφωνίε. Και εγώ ειλικρινώς σα λέω ότι θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο και θα πρέπει με εκβιασμούς να σε εκβιασμούς να απαντάμε με εκβιασμού. Η κυρία Ρόντουστ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώς ε, δεν με λάβατε υπόψη, αλλά έτσι είναι πιο εύκολη κατάσταση για μένα γιατί δεν χρειάζεται ε, ε, να επαναλάβω ορισμένα πράγματα καθότι στηρίζω όλα τα σχόλια και πρέπει να πω ότι η εργασία αυτή ήταν πολύ σωστή η οποία απέδειξε ότι αυτό το οποίο επιθυμούμε από μία συμφωνία, μία κατάσταση η οποία θα είναι επικερδής για όλα τα μέλη δεν είναι δεδομένη. Δεν θα αναφερθώ μόνο στο θέμα της Σπυραλίευσεως, αλλά ήδη εκεί ε, θα είχαμε αμέσως μία αρνητική αξιολόγηση της συμφωνίας και γι' αυτό ε, αναρωτιέμαι αν δεν θα μπορούσαμε από κοινού να χρησιμοποιήσουμε την καλή πείρα που είχαμε για την Μαυρικανία μέσω του ψηφίσματος να τη χρησιμοποιήσουμε και για το Μαρόκο. Να πούμε δηλαδή πώς εμείς φανταζόμαστε μία μελλοντική ε, συμφωνία τι επιθυμούμε να περιλαμβάνεται σαν ρήτρε και ε, τι μπορούμε να αποδεχτούμε. Νομίζω ότι αυτό είναι λογικό και πρέπει να κινηθούμε αμέσως διότι ο χρόνος περνά. Τους τελευταίους μήνες προσπάθησαμε να λάβουμε ε, υλικό από όλες τις πλευρές. Όταν κοιτάζω όμως την έκθεση Χάγκλουν πρέπει να πω ότι πολλά θέματα κρεμούν ακόμη, δεν έχουν απαντηθεί και ε, ναι μεν η κυβέρνησή μου έχει αποδεχθεί τη συμφωνία γιατί θεωρεί ότι άλλαξε η κατάσταση αλλά ο κύριος Χάγλουν πολύ σωστά απέδειξε ότι δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε αυτή την συμφωνία με στην παρούσα της μορφή και θα πρέπει Φεβρουαρίου να έχουμε ε, μέσω ενός ψηφίσματος μία κατάσταση την οποία όλοι μπορούμε να αποδεχθούμε. Ε, παρακαλώ αυτά να τα σημειώσετε γιατί νομίζω ότι ότι πρόκειται για βασικά θέματα. Κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο. Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω ορισμένα στοιχεία σχετικά με τα όσα ελέγχθησαν σήμερα το πρωί. Καταρχήν να διαβεβαιώσω όσους μας ακούν επί των διαδικασιών διότι οι διαδικασίες όντως έγιναν σεβαστές. Ναι μεν επιταχύναμε το ρυθμό, υπήρχε ένα πρωτόκολλο που και ανανεώθηκε ε, για ένα έτος αλλά σεβαστήκαμε τα δικαιώματα όλων των θεσμικών οργάνων. Όσον αφορά την έκθεση αξιολογήσεως θα ήθελα να σας πω ότι η έκθεση αυτή είναι ένα έγγραφο εργασίας ε, που έχει συνταχθεί σε μία γλώσσα εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν είναι μία αξιολόγηση της ιδίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι στοιχεία που πρέπει να θυμάστε. Ενδεχομένως αργήσαμε να παρουσιάσουμε μία αγγλική μετάφραση. Πρέπει να σας πούμε ότι συνήθως οι εκθέσεις αυτές δεν μεταφράζονται και μόνο κατ' εξαίρεση δεχθήκαμε παρόλη την φύση και το χαρακτήρα αυτών των εγγράφων να το μεταφράσουμε. Δηλαδή υπομαλά συνθήκας δεν επρόκειται να υπάρξει μετάφραση. Ίσως ε, το Κοινοβούλιο θα μπορούσε μέσω των υπηρεσιών του να έχει μεταφράσει πιο γρήγορα το κείμενο αυτό διότι πρόκειται για ένα εκτενές κείμενο. Ε, μας βοηθά όμως στην φάση αξιολογήσεως το έγγραφο αυτό χωρίς να αντικατοπτρίζει τις απόψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να αποστασιοποιηθούμε και να το θυμόμαστε αυτό. Ε, όντως τελικά πρόκειται για ένα θέμα που είναι ίσως λιγότερο ενδιαφέρον για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε ε, και είναι αντίθετο αλλά πρέπει να πούμε ότι δύο από αυτές τις κατηγορίες υποχρησιμοποιούνται. Πρόκειται δηλαδή για τα βυθικά είδη τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ελάχιστα στα πλαίσια της συμφωνίας. Πρόκειται όμως για ένα έγγραφο το οποίο παρέτεινε την προηγούμενη συμφωνία προσπαθώντας να έχουμε μια πιο εποφελή οικονομική και εμπορική συμφωνία. Χρειάζεται να βαθύνουμε τα ε, στοιχεία τα επιστημονικά ε, και υπάρχουν ορισμένες αμφιβολίες ε, θα πρέπει να υπάρχει μία σωστή και ποιοτική επιστημονική αξιολόγηση της εκθέσεως και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα συγκαλέσουμε μία κοινή επιστημονική επιτροπή μαζί με τις μαροκινές αρχές για να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα θέματα και την ε, κατάσταση των αλλιευμάτων και θα συνέλθει η Επιτροπή αυτή τον Οκτώβριο. Αναφερθήκατε στον τομέα της αλληλείας στο Μαρόκο. Έχουμε λάβει στοιχεία τα οποία μας έδωσε το Μαρόκο και τα μεταφέραμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προέβημεν σε μια συνθετική εργασία και πρέπει να πούμε ότι όλοι εποφελούνται υπάρχει μια θετική αξιολόγηση ε, και ε, επιρροή σε ολόκληρο το Μαρόκο και με τις μεροκινές αρχές ε, αξιολογήσαμε ε, τις ε, τομεακές ε, πρόοδους που έχουν γίνει σχετικά με τα σειρώμενα εργαλεία που είναι σημαντικά για το περιβάλλον, για την οργάνωση των λιμένων, για τις επαγγελματικές οργανώσεις. Υπάρχουν πολλές δράσεις που χρηματοδοτούνται και παρακολουθούνται εκ του σύνεγγις όσον αφορά την πρόοδό τους έχουμε και κοινέ συζητήσεις και ε, ε, ε, αποβιβάσεις σχετικά με ορισμένα αλλιεύματα και ο, πολύ σωστά ο κύριος Στίβενσον αναφέρθηκε στις αποβιβάσεις στο Ντακάρ ορισμένων αλλιευμάτων από την περιοχή της Δυτικής Σαχάρας. Θα ήθελα τώρα να επανέλθω εις το εδαφικό χαρακτήρα της συμφωνίας αυτής που κατά τη γνώμη μας συνάδει με το διεθνές δίκαιο και ε, βλέπουμε ε, τις επιπτώσεις στην περιοχή της Δυτικής Σαχάρας γι' αυτό και περιλάβαμε ένα νέο και ουσιαστικό άρθρο το 7.4 μέσω του πρωτοκόλλου και θέλω να σας τονίσω το άρθρο αυτό διότι συμφώνησαν οι Μαροκινοί για να παρουσιάζεται δηλαδή να υπάρχει μία έκθεση την οποία θα υποβάλει το Μαρόκο ένα μήνα πριν από την εκπνοή του πρωτοκόλλου σχετικά με τις επιπτώσεις τις οικονομικές και τις εμπορικές που περιμένουμε από συμφωνία αυτή και να τις αξιολογήσουμε σύμφωνα με το άρθρο αυτό το 7.4. Ε, λοιπόν, έτσι έχουμε ένα νομικό τρόπο να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν ισοσκελισμένες συνέπειες της συμφωνίας αυτές σε όλο το έδαφος ε, και την επικράτεια της ε, χώρας. Η κυρία Φράγκα ερώτησε τι θα γίνει σχετικά με τη στρατηγική μετά τις 27 Φεβρουαρίου αλλά δεν είμαι εξουσιοδοτημένος να σχολιάσω το θέμα αυτό το οποίο θέλει ακόμη σκέψη και συζήτηση ε, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον αυτού του πρωτοκόλου και όσον αφορά τα άλλα θέματα τα οποία ανθίξαμε, δυστυχώς ε, κυρία Λέβιν πρέπει να πω ότι ε, δεν ε, είμαι αρμόδιος για να, το, να απαντήσω στο ερώτημα αυτό. Ευχαριστώ. Ναι, ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, ε, εφόσον το ξέχασα, ευχαριστώ ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή την κίνηση καλής θέλησης, να μεταφράσει δηλαδή την ε, έκθεσή της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από ό,τι καταλαβαίνω και πάλι, θεωρούν ότι δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε κάποια επίσημα πράγματα για να εξηγήσουμε για ποιο λόγο ε, έχει όπως έχει ε, η διαδικασία. Αυτό όμως δεν αλλάζει την ε, πολιτική πραγματικότητα που βλέπει το Κοινοβούλιο ότι δηλαδή ήταν χειριστός ο χειρισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να το έχουμε κατά νου. Σχετικά με το feedback που μου δώσατε, σας ευχαριστώ. με τη συζήτηση που έγινε φαίνεται ότι πόσο σημαντικό είναι αυτό το ζήτημα, πόσο πολυδιάστατο. Ε, στρέφομαι προς τον συνάδελφο Καντέ και άλλους ε, που είπαν ότι το Μαρόκο είναι ένας ε, σημαντικός εμπορικός εταίρος. Κοιτάξτε, από κοινού θα το αξιολογήσουμε αυτό, συμφωνώ μαζί σας, πως το Μαρόκο είναι σημαντικός εμπορικός εταίρος ε, για την Ένωση στο σύνολό της και μεμονωμένα για κάποια κράτη-μέλη. Άρα είναι ευαίσθητο, λεπτό και σημαντικό το ζήτημα, όμως αυτό δεν αλλάζει τίποτα στα στοιχεία της θέσης αξιολόγησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωραία, ζυγίσουμε τι είναι πιο σημαντικό. Ε, αυτά που θέλουν ο Κάντε και άλλοι να τονίσουν ε, και για, ο λόγος δηλαδή για τον οποίο πολλές χώρες υποστηρίζουν αυτή τη συμφωνία και ούτω καθεξής. Ναι, ισχύει και αυτό. Ε, ελπίζω αυτό να γίνεται για πολιτικούς λόγους και να μην ε, προφασιστείτε τη λογική γιατί δεν ισχύει αν αναλύσετε την έκθεση αξιολόγηση. Στην αρχική μου παρουσίαση σήμερα δεν ερμήνευσα οτιδήποτε, παρέθεσα τμήματα, ε, αποσπάσματα της έκθεσης. Δεν είναι η δική μου άποψη αυτή την οποία ακούσατε. Είναι η έκθεση της Επιτροπής και ήθελα να τονίσω ότι αυτά είναι ε, γεγονότα αντικειμενικά. Ελπίζω που συμπεριλαμβάνονται μέσα σε αυτή την έκθεση αξιολόγηση. Δεν έχουν διαβάσει πολλοί συναδελφοί ε, αυτή την έκθεση. Περισσότεροι όμως έχουν σχόλια και απόψεις. Συγγνώμη, αλλά όταν έχετε αμφιβολίες, σας παραπέμπω σε αυτές τις εκθέσεις. Θα σας το δώσει την έκθεση η γραμματεία. Πάρτε τη μαζί σας, μπορείτε να τη φωτοτυπήσετε ή πηγαίνετε στη γραμματεία ε, και διαβάστε τη. Όπως είπε και η κυρία Φράγκα, δεν είναι το πιο ευανάγνωστο κείμενο που υπάρχει, αλλά πρέπει να το διαβάσετε για να δείτε και να διαπιστώσετε η διεισόμαση ότι αυτά που ακούσατε από το στόμα μου δεν είναι δικέ μου απόψεις αλλά είναι στοιχεία από την έκθεση. Ε, βασίζομαι στην έκθεση πρόκειται για γεγονότα, αδιαμφισβήτητα. Ε, για τη Δυτική Σαχάρα εγώ προσωπικά είμαι πεπισμένος πως ε, επί τη βάση των πληροφοριών που λάβαμε από το συναδέλφους όπως ο κύριος Στίβενσον αλλά και από τις ε, καρποφόρες συζητήσεις με τις, Μαρό, ε, αρχές του Μαρόκου και παρεμπιπτόντως να πω ότι ήταν αγαστή η συνεργασία, μας βοήθησαν οι αρχές του Μαρόκου, ε, μας έδωσαν τις πληροφορίες που ζητήσαμε. Λοιπόν, σε σχέση με όλα αυτά τα σχόλια, καλό θα ήταν να λάβουμε υπόψη και αυτή την πλευρά. Πάντως, πληροφορίες που έχω στη διάθεσή μου αποδεικνύουν ότι όντως δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης με τη συμφωνία, όντως βελτιώνεται η οικονομική κατάσταση, αλλά μπορούμε να δούμε σε ποιο βαθμό βελτιώνεται ε, η κατάσταση σε σχέση με τα αρνητικά στοιχεία, γιατί είναι συγκεκριμένη και η διατύπωση με στην έκθεση αξιολόγηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει στοιχεία σε σχέση με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου για την κλαδική υποστήριξη. Αναφέρει σαφέστατα η έκθεση αξιολόγηση ότι ε, η υποστήριξη στον κλάδο από πλευρά τη Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή ε, δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Δεν, έχει, δεν έχουν διοχετευθεί αυτά τα κονδύλια στον κλάδο. Αν θυμάμαι καλά, ένα λεπτάκι. Μόνο 21 από 54 εκατομμύρια που έπρεπε να διοχετευθούν στον κλάδο τελικά πήγαν, έφτασαν στον προορισμό τους, αν θυμάμαι καλά λιγότερα από τα μισά δηλαδή κονδύλια που προορίζονταν για τη στήριξη του κλάδου. Οπότε θα πρέπει να σημειωθεί κάποιος κάποια πρόοδος. Εντυπωσιάστηκα με τις βελτιώσεις που επέφερε το Μαρόκο στον αλλιευτικό κλάδο. Είναι σημαντικό να το πούμε και αυτό. Αλλά πρέπει ταυτόχρονα να πούμε ότι δεν έγινε αυτό χάρη στην πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά χάρη ε, στους ε, πόρους ε, που έχει το Μαρόκο, χάρη στην εθνική στρατηγική. Ε, δεν ε, έχουμε τόσο μεγάλο ρόλο ως Ευρωπαϊκή Ένωση και πάλι τώρα βασίζομαι σε στοιχεία της έκθεσης για να το ισχυριστώ αυτό. Και πάλι για τη Δυτική Σαχάρα νομίζω θα ήταν συνετό από ε, πολιτικής σκοπιάς να τονίσουμε ότι η συμφωνία με το Μαρόκο επηρεάζει θετικά τη Δυτική Σαχάρα. Ωραία. Αλλά υπάρχει και η πολιτική διάσταση του ζητήματος. Δηλαδή η συμφωνία αυτή είναι νομικά έγκυρη όταν μιλάμε για τη Δυτική Σαχάρα. Ο συνάδελφος ε, Ρουέντα ε, ε, εξέφρασε την άποψή του και δεν μου αρέσει όλη αυτή η συζήτηση γιατί επικρατεί σύγχυση. Νομίζω ότι θα πρέπει ίσως να διαχωρίσουμε αυτά που πραγματεύεται αυτός μέσα στην έκθεσή του και τα στοιχεία που απασχολούν εμένα για να είναι σαφέστερη η συζήτηση. Πρόεδρε, ε, όπως είπα, ε, προτρέπω τους συναδέλφους να μελετήσουν αυτή την έκθεση. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα τα στοιχεία και με τα χαράς να τα ξανασυζητήσουμε. Ε, στη συνεδρίασή μας τον Οκτώβρη γιατί πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και τέλος για τη μελλοντική στρατηγική με ερώτηση κυρία Φράγκα. Ε, δε, δυστυχώς δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχει εντολή για να τοποθετηθεί μου λέει. Ε, ωραία. Άρα και εγώ δεν έχω ιδέα για τις προθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μήπως ε, ε, ξεχνάτε ότι πριν από ένα χρόνο προσπαθήσαμε όλοι να μάθουμε τι γίνεται και πήραμε διαφορετικές απαντήσεις και τελικά τι μάθαμε, ότι παρατάθηκε η ίσχυση του πρωτοκόλλου ε, και πολύ φοβάμαι θα επαναληφθεί αυτό το σενάριο και ε, σοβαρευτείτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλώ γιατί δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Να σας ενημερώσω απλώς για το χρονοδιάγραμμα. Παρουσίαση θα έχουμε τον Οκτώβριο, ψηφοφορία στις 22 Νοεμβρίου και ε, κατά πάσα πιθανότητα θα ψηφιστεί στη συνέχεια στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Ευχαριστούμε τον κύριο Χάγλουντ ε, και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ολοκληρώθηκε και αυτό το σημείο. Το σημείο 8 έχει αναβληθεί. Στο σημείο 9 τώρα της ημερήσιας διάταξης έχουμε την υιοθέτηση για το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων για το 2012 Δεν υπήρξε καμία ένσταση για το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, επομένως θεωρούμε ότι εγκρίνεται. Και με αυτό ε, έχουμε ολοκληρώσει και το ε, σημείο 9. Το 10 το συζητήσαμε. Υπάρχει τίποτα από τα διάφορα. Εμείς δεν έχουμε. Αν θέλετε μπορείτε να το θέσετε εσείς. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 19 Σεπτεμβρίου στις 3 το απόγευμα εδώ στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ σε όλους. Πέρα συνεδρία.